Γεια σας ε, συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ο χρόνος πιέζει, οπότε θα ήθελα να κηρύξω την άνοιξη της ε, δεύτερης συνάντησης της Επιτροπής, Εξεταστικής Επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, ε, που είναι όμως η πρώτη πραγματική ουσιαστική συνάντηση. Αν δεν έχετε σχόλια για την ημερήσια διάταξη, την υιοθετούμε χωρίς αλλαγές. Υπάρχει διερμηνία σε 18 γλώσσες. Μία από αυτές είναι τα δανέζικα. Ε, η συνεδρίαση μεταδίδεται από το ίντερνετ και γίνεται χωρίς ε, ε, αντίγραφα των εγγράφων σε χαρτί. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 28 Απριλίου και θα καλέσουμε εκεί έχουμε καλέσει και θα έρθουν ο κ. Dirk Ποστέλς από την Ένωση Ελέγχου Εκπομπών με Καταλήτη και ο κ. Ούντο Λάμπρεχτ του Ινστιτούτου για την Ενέργεια για την Περιβαλλοντική Έρευνα της Χαϊδελβέργη. Έχουμε προετοιμάσει ένα γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο θα σταλεί στις εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι δηλαδή τα αρμόδια υπουργεία και στις ε, υπηρεσίες έγκρισης τύπου. Του ζητήσαμε να μας στείλουν τις απαντήσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου. Θα δούμε αν αυτό είναι δυνατόν. Έτσι ώστε να έχουμε αρκετό υλικό για να διαβάζουμε κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών μας. Επίσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ζητήσει διάφορα πράγματα, μεταξύ αυτών και τη σύσταση και τα πρακτικά ε, διαφόρων ομάδων πυρογνωμόνων, καθώς επίσης και την αλληλογραφία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής με διάφορες ενώσεις, ε, οργανισμούς κλπ. Τέλος, θα δημοσιευθεί ένα, μια διεύθυνση αλλογρα... ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο site μας έτσι ώστε να μπορεί οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία να μας στείλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Αν δεν υπάρχουν σχόλια θα ήθελα να περάσω στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης και να ξεκινήσουμε και την πρώτη πραγματική ακρόαση ε, της μέρας και της Επιτροπής μας. Καλωσορίζω την κυρία Ντελιλά Αλ Κουντάιρη έτσι διαβάζετε το όνομά σα. Ωραία. Διευθύντρια και τον κύριο Αλουά Αλόης Κράσενμπρινκ, επικεφαλής ε, της ε, μονάδας ε, βιώσιμων μεταφορών του κέντρου, Κοινού Κέντρου Έρευνας. Έχουμε στη διάθεσή μας μια ώρα και 40 λεπτά για αυτή την ακρόαση. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχετε λάβει τις απαντήσεις σε ένα πρώτο ερωτηματολόγιο που είχαμε στείλει στο JRC, στο Κοινό Κέντρο Έρευνας. Ελπίζω να τις διαβάσατε. Δεν χρειάζεται να ξαναθέσουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Θα τις χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να εμβαθύνουμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αλκουντάιρη. Παρακαλώ πολύ, μια εισαγωγική παρέμβαση, το πολύ 10 λεπτά και μετά θα σας ξαναδώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε, Αντιπρόεδροι, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ε, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας εξηγήσω το ρόλο και, την εργασία, και το έργο του JRC, του Κοινού Κέντρου Έρευνας, σε σχέση με την νομοθεσία για τις εκπομπές ε, οχημάτων. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω τι έχουμε κάνει για να ε, μειώσουμε το, τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές μετρήσεις, μετρήσεις σε πραγματική χρήση και τις μετρήσεις των, ε, που γίνονται στα εργαστήρια. Μετά θα σας πω τι έρευνα έχουμε κάνει για τις πραγματικές εκπομπές ε, και πώς αυτές ε, τις ε, κοινοποίησαμε στην Κομισιόν και στους άλλους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω τις τα τεχνικά προβλήματα, τις δυσχέρειες που έχουμε στην εισαγωγή αυτού αυτής της μεθόδου των πραγματικών εκπομπών στην διαδικασία έγκρισης τύπου και τέλος θα σας πω πώς στηρίζουμε το καινούριο πλαίσιο ε, έγκρισης τύπου. Κατρίνη, σας εξηγήσω ποιο είναι ο ρόλος μας Είμαστε η Υπηρεσία Έρευνας ε, και Γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μας δίδεται εντολή, παίρνουμε και δική μας πρωτοβουλία, να παρέχουμε επιστημονικές ε, ε, συμβουλές στην, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, οι εκπομπές των αυτοκινήτων είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς εργαζόμαστε με κατόπιν εντολής από κάποιον που σχεδιάζει μια καινούργια πολιτική είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε εκτός και στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, δεν είχαμε εντολή να ελέγξουμε τη συμμόρφωση ή την έγκριση τύπου ε, των κέρνουριων αυτοκινήτων που έμπαιναν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιθέτως να αναπτύξουμε μεθοδολογίες δοκιμών ελέγχου. Ε, τα αποτελέσματά μας ε, λαμβάνονται σε, σε εγκαταστάσεις μας που είναι υπερσύγχρονες και ε, κοινοποιούνται στις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG Grow που ήταν παλιότερα DG Επιχειρήσεων, DG Κλίμα και DG Env περιβάλλοντος. Ιδιαίτερως για να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν καινούργια ε, ε, νομοθεσία για τις ε, οριακές εκπομπές, ρήπων και εκπομπών. Επίσης, ε, για να καθοριστούν στόχοι για την ε, κατανάλωση ε, καυσίμων, διοξιδίου του άνθρακα κλπ. και για να συμμετέχουμε στην, ε, ε, στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, ε, τις τεχνολογίες που έχουν σχέση με την οικολογία και την καινοτομία. Τώρα, ο στόχος της εργασίας μας για τα, τις πραγματικές εκπομπές ξεκινήσαμε το 2011 αυτή τη διαδικασία. Το βασικό ζήτημα ήταν πόσο ε, αντιπροσωπευτικά ή αντιπροσωπευτικέ ήταν οι δοκιμές έγκρισης τύπου ε, σε σύγκριση με τις εκπομπές που θα μετρούσε κανείς σε πραγματικές συνθήκες. Με άλλα λόγια, σε ποιο βαθμό οι μετρήσεις που γίνονται στα εργαστήρια αντιπροσωπεύουν και ελέγχουν επαρκώς ε, τις πραγματικές εκπομπές. Και αν υπάρχει μεγάλη διαφορά, ποια θα ήταν η μεθοδολογία για να μειωθεί αυτή. Ε, για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα χρειάζεται πραγματικά πολλή έρευνα, ε, μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες ε, και την χρήση, ανάπτυξη και χρήση φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών που ονομάζονται PEMS με τα αγγλικά αρχικά τους. Εμείς ξεκινήσαμε από το 2000, είχαμε ξεκινήσει ήδη την διαδικασία έρευνας για τέτοιου μετρήσεις, ακόμα και πριν το 2011. Ξεκινήσαμε ε, από το 2004 συγκεκριμένα. Όμως ε, τότε είχαμε εστιάσει όχι σε ελαφρά οχήματα, αλλά σε ε, βαρέα οχήματα και τη μέτρηση των πραγματικών εκπομπών, εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, λεωφορεία, φορτηγά και τέτοια. Μετά από εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, ξεκινήσαμε μια, ένα πρόγραμμα, συνεργατικό ερευνητικό πρόγραμμα, ε, για να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία και μια αναλυτική μέθοδο για να ε, δούμε το κατά πόσον τα βαρέα οχήματα συμμορφώνονται σε ό,τι αφορά τις εκπομπές τους με τις απαιτήσει της νομοθεσίας ε, και κατά πόσον αυτό τα αποτελέσματα συμπίπτουν με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου. Εκείνη την εποχή ε, τα φορητά συστήματα μέτρηση ήταν σχετικά καινούρια. Υπήρχε μόνο ένα σύστημα που ήταν εμπορικά διαθέσιμο και ήταν ε, βαρύ, δύσκριστο ε, και, και ενεργοβόρο. Για βαρέα οχήματα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά όχι για ελαφρά οχήματα. Το 2007 το JRC έκανε τις πρώτες προσπάθειες να λειτουργήσει PEMS και σε ελαφρότερα οχήματα ξεκινήσαμε με ένα διαρευνητικό ερευνητικό πρόγραμμα για να διαπιστώσουμε το κατά πόσον υπάρχουν ε, διαφορέ ανάμεσα στι εκπομπέ που υπολογίζονται στο εργαστήριο με τι πραγματικέ εκπομπέ και να δημιουργήσουμε μια, να αναπτύξουμε μια μεθοδολογική προσέγγιση για ε, επιβατικά οχήματα. Διαλέξαμε 12 οχήματα από μια επιχείρηση ενοικίαση αυτοκινήτων προσπαθώντα να καλύψουμε όλου του τύπου μηχανών, ε, βενζίνης, δίζελ ε, και προδιαγραφών εκπομπών Euro 3, 4 και 5. Βασιστήκαμε στο, στις διάφορες ε, τεχνολογίες μηχανών, μεγέθη κλπ. ανεξαρτήτως ε, μάρκας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα εκπομπές διοξιδίων, ε, του αζότου ε, με, σε αυτοκίνητα diesel Euro 3 ως 5 ξεπερνούσαν κατά 4 έως 7 φορές τα όρια και για συγκεκριμένα μοντέλα μέχρι και 14 φορές. Αυτά τα αποτελέσματα, χωρίς όμως συγκεκριμένη αναφορά σε μοντέλα, ε, κοινοποιήθηκαν στην Κομισιόν η οποία συγκάλεσε, ε, ε, διοργάνωσε ένα τεχνικό εργαστήρι στις 23 Νοεμβρίου 2010 με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν αυτά τα πράγματα και το τι σήμαιναν στην πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί τη βάση των συζητήσεων αυτών, η Κομισιόν αποφάσισε να συστήσει μια τεχνική ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη ε, δοκιμασιών σε πραγματικές συνθήκες, ε, δοκιμών συγγνώμη, σε πραγματικές συνθήκες. Το 2001 αυτά τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν ε, κιόλας ε, σε επιστημονικό άρθρο και μάλιστα η αποδοχή του αποδεικνύει ότι ήταν και βάσιμα. Από τη στην αρχή του 2011 η ομάδα εργασίας για τις κομπές σε πραγματικές συνθήκες για ελαφρά οχήματα, RDE-LDV έτσι ονομάζονταν, ε, δημιουργήθηκε από την Κομισιόν με συμμετοχή των κρατών μελών, ε, της αυτοκινητοβιομηχανία, ε, ε, εμπειρογνωμόνων μη κυβερνητικών οργανώσεων και εμπειρογνωμόνων τη Κομισιόν. Επιπλέον, εκτό των PEMS, ε, αναλύθηκαν και άλλε τρει μέθοδοι μέτρηση πραγματικών εκπομπών. για παράδειγμα, χρήση το, τον, του, πολλαπλών κύκλων δοκιμών, όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Δεύτερον, ε, η χρήση του τυχαίων ε, δοκιμών ε, κύκλου σε εργαστήριο και τρίτον μοντελοποίηση, πράγμα όμως που δεν του δώσαμε μεγάλη σημασία διότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εφικτό να γίνει μοντελοποίηση. Η Κομισιόν το 2012 ζήτησε από το JRC μια επιπλέον μελέτη για να διαπιστώσουμε το κατά πόσον αυτές οι μέθοδοι ήταν τεχνικά βιώσιμες ε, και για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για τις πραγματικές ε, εκπομπές και τις πραγματικές συνθήκες ε, λειτουργίας των ελαφρών οχημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα PEMS θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για ελαφρά οχήματα υπό προϋποθέσεις. Το 2013 το, τα αποτελέσματά μας υποβλήθηκαν στην ομάδα εργασίας RDLDV και δημοσιεύθηκαν στη δεύτερη έκθεση που ε, δημοσίευσαμε για αυτές τις διαδικασίες. Κατόπιν αυτών, η ομάδα εργασίας ε, αποφάσισε να, κρατήσει, να διατηρήσει τα πέμψο στην προτιμόμενη μέθοδο εργασίας. Τα επόμενα δύο χρόνια αναπτύξαμε δύο μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγηση δεδομένων για τη στατική αισθητική ανάλυση των μετρήσεων με PEMS. Ε, η ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων από μια ομάδα εργασίας όπως η RD ή η LDV ε, ήταν πολύ σημαντική για να εξασφαλίσουμε ε, την συμμόρφωση με τα, με τις, όρια εκπομπών. Τώρα, στην πρότασή μας για την αναθεώρηση του σχεδίου του ε, πλαισίου ε, έγκρισης τύπου, η Κομισιόν πρότεινε μεταξύ άλλων μέτρων ε, να ενισχύσουμε την ανεξάρτησία των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου ε, με νέες διατάξεις έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα οχήματα θα συμμορφώνται πραγματικά με την νομοθεσία. Για παράδειγμα ένα μηχανισμό peer review, ε, αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων ε, για τις τεχνικές υπηρεσίε και τη δυνατότητα να γίνονται δοκιμές από αυτοκίνητα, σε αυτοκίνητα της αγοράς όχι μόνο στο εργαστήριο. για να εγκριθεί αυτή η πρόταση, θα πρέπει το JRC να είναι η υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για την ε, εφαρμογή αυτών των, ε, την υλοποίηση αυτών των ε, μετρήσεων στην νέα νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να γίνεται δυνατή η δοκιμή με μεθόδους που δεν είναι στάνταρ μέχρι τώρα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις παράκαμψης, γνωρίζουμε τη δυνατότητα χρήσης τους. Δεν γνωρίζουμε όμως αν κάποια από τα αυτοκίνητα τα οποία εμείς δοκιμάσαμε ε, είχαν τέτοιου είδου ε, διατάξεις το 2007-2010. Ε, δεν το είχαμε λάβει υπόψη μας αυτό στην τότε έρευνα μας. I think. I would like to just end basically... Θα ήθελα τέλος να προσθέσω α, θα, ε, συμπερασματικά ότι πω, να πω, επαναλάβω ότι το JRC ως υπηρεσία έρευνας και επιστήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να βρίσκεται ε, στο επικεφαλής της εργασίας που στηρίζει τις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές μείωσης των εκπομπών στο αυτοκίνητο βιομηχανία και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πλήρη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Το και σας περιμένουμε τον Ιούλιο στα εργαστηριά μας. Πρόεδρος, ναι, και εμείς το περιμένουμε. Συνάδελφοι, έχουμε μια μισή ώρα. Έχουμε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο ε, πέντε λεφτά, ε, με ερωτήσει το πολύ ένα λεπτό και μια απάντηση μετά. Το, ο βουλευτής που κάνει την ερώτηση μπορεί να σταματήσει τον ομιλητή, με φιλικό τρόπο θα έλεγα, και να κάνει μια ερώτηση, χωρίς όμως να παρατείνουμε το πεντάλεπτο. Στο δεύτερο γύρο Αντί για πέντε λεπτά θα έχουμε τρία λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με το συζητητή μας, ο κ. Ε, Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτέλους ξεκινάμε ε, την πραγματική μας ακρόαση. Ευχαριστώ την κυρία Αλκουντέρα που ήρθε εδώ. Έχω δύο βασικές ερωτήσεις. Πρώτον, Και στις εκθέσεις του 11 και του 13 το κέντρο βρήκε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις εκπομπές ε, μετρημένες στο εργαστήριο και τις πραγματικές εκπομπές. Κατά την οδήγηση δηλαδή. Και στην ε, απάντηση 3α στο ερωτηματολόγιο λέτε ότι δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι υπήρχαν στρατηγικές νόμιμες για την αλλίωση των αποτελεσμάτων Και η έρευνα ε, για το θέμα αυτό δεν ήταν στο πλαίσιο των εργασιών του ερευνητικού κέντρου. Γιατί όχι. Γιατί ε, θέλατε να αναπτυχθούν νέες δοκιμές. Αλλά δεν ξέρατε ποιε ήταν, ποιες ήταν οι δυναμίες των παλιών δοκιμών, έτσι. η ερώτησή μου είναι γιατί δεν υπήρχε αυτό στο πλαίσιο των εργασιών σας. Και εσείς το, ως κέντρο ζητήσατε ε, από την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο των εργασιών σας για να ασχοληθείτε και με τις συσκευές αλλίωσης. Ε, από την πρώτη συνεδρίαση του RDV-LDV της Ομάδας Εργασίας, φανταστικός τίτλος, 31 Ιανουαρίου του 2011 που ασχολιόταν ακριβώς με την ανάπτυξη νέων συμπληρωματικών διαδικασιών δοκιμών και δύο χρόνια μετά, όπου επιτέλους μία από τις τέσσερις επιλογές επε, ε, επελέγει, ας πούμε. Γιατί χρειαστήκατε δύο ολόκληρα χρόνια για να επιλέξετε ανάμεσα αυτές τις τέσσερις εναλλακτικές λύσεις που είχατε. Let me Γιατί υπήρχαν αυτές τεράστιες ε, διαφορές ε, ανάμεσα στα εργαστηριακά αποτελέσματα και στις πραγματικές μετρήσεις. Οι διαφορές υπάρχουν λόγω του ότι έχουμε άλλες τελείως συνθήκες, συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Γι' αυτό η Κομισιόν ζήτησε από το κέντρο να κάνει ακριβώ αυτή την ε, έρευνα, γιατί ξέραμε τότε ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα ή μάλλον οι εργαστηριακές δοκιμές δεν μπορούν να προσωμιώσουν, ας πούμε, να πλησιάσουν ε, τις πραγματικές συνθήκες λόγω του ότι υπάρχει ο καιρός, υπάρχει το θέμα της ταχύτητας, υπάρχουν διάφορες παράμετροι, πούμε, που δεν μπορούν να προσωμιωθούν. Και επομένως οι πραγματικές εκπομπές αντανακλούν και δείχνουν την ανεπάρκεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Δεν ε, είδαμε να έχουμε τρομερά προβλήματα στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, βενζινοκίνητα όσο στα ντίζελοκίνητα αυτοκίνητα και κινητήρες. Ε, στο 2007, ε, κάθετος 6, κάθετος 15, υπήρχε η εντολή ε, η Κομισιόν να βελτιώσει τις διαδικασίες δοκιμών, ούτως ώστε να μειωθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα στις ε, εργαστηριακές και στις πραγματικές δοκιμές. Τα ξέραμε τότε ότι αυτό το κενό, αυτή η διαφορά υπήρχε και θέλαμε να βελτιώσουμε τότε τις εργαστηριακές δοκιμές θέλαμε να δούμε τι επιτυχίες είχαμε στα βαριά οχήματα, τόσο ώστε να προσαρμόσουμε το φορητό σύστημα εκπομπών και να το χρησιμοποιήσουμε και στα ελαφρά οχήματα, για να δούμε ε, μήπως με τη χρήση των PEMS θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτή τη ε, διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στις εργαστηρια, στα εργαστηριακά αποτελέσματα και στις, ε, στα πραγματικά. Μας είπατε, με ρωτάτε γιατί δεν ε, εξετάζαμε τότε και αυτές τις συσκευές αλλίως των αποτελεσμάτων. Από το τέλος της δεκαετίας του 90 ξέραμε ότι υπήρχαν τέτοιες ε, δυνατότητες να αλλοιώσουμε τα αποτελέσματα μέσω διαφόρων συσκευών, ας πούμε. Γι' αυτό υπάρχει και ένα άρθρο στον ε, κανονισμό του 2007, τον 615, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Για να τα ανοιχνεύσουμε όμως αυτά τα συστήματα, αυτές τις συσκευές, θα πρέπει οι διαδικασίες δοκιμών να σχεδιαστούν με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να μην έχουμε την προσέγγιση έγκριση τύπου που είχαμε. Το βασικό είναι να συμπληρώνουμε με, πραγμα... με μετρήσεις των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή κατά διάρκεια της οδήγησης, και να συμπληρώνουμε τις εργαστηριακές δοκιμές. Σε εκείνη τη φάση όμως, το... στο παρελθόν, δεν Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγκριση για να ανοιχνεύσουμε αυτές τις συσκευέ. Γιατί το βασικό ήταν ε, να εφαρμόσουμε την εντολή της Κομισιόν, να βελτιώσουμε δηλαδή το επίπεδο της πρόληψης, τους ελέγχους και τη μείωση των εκπομπών όλων των ειδών οχημάτων. Να διακόψω, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Αλλά από την άλλη, είδαμε ότι η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα των εργαστηρίων και των πραγματικών εκπομπών αυξάνονται. Δεν σας έκανε εντύπωση γιατί συνέβαινε αυτό. Είπατε ήδη ότι η χρήση τέτοιων συσκευών αλλίωσης ήταν κάτι γνωστό, δεν ήταν καινούριο. Ήδη από την δεκαετία του 90. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να επεκτείνετε το πεδίο εφαρμογή είτε από μόνοι σα, α πούμε, αυτεπάγγελτε, είτε να το ζητήσετε ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ζητήσατε να σα δοθούν περισσότεροι πόροι για να κάνετε αυτή την έρευνα. Απλή ερώτηση, ναι ή όχι. Δεν είχαμε την εντολή, λέει η Διευθύντρια, σε επίπεδο εντολής. Ποτέ δεν ρωτήσατε. Ποτέ δεν ρωτήσατε την Κομισιόν, μπορείτε να μα δώσετε αυτή την εντολή. Όχι, όχι, δεν υπήρχε ποτέ η υποψία ότι οι διαφορές που βλέπαμε οφειλόταν στην ύπαρξη αυτών των συσκευών αλλίωση. Τυφλοί ήμασταν, αν θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Θέλαμε απλώς ε, τα φορητά συστήματα μέτρηση των εκπομπών να τα χρησιμοποιήσουμε σε περισσότερα οχήματα, σε περισσότερα ίδια οχημάτων και να συμπληρώσουμε έτσι τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ για να συνεργαστείτε μαζί μας. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο, κύριος, ο προηγούμενος ομιλητής. Εσείς είχατε στοιχεία, στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία, το τονίζω. Όχι απλώς υποψίες για, αυτά για αυτές τις ε, συσκευές αλλίωσης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Αν ναι, αν είχατε τέτοια στοιχεία, τι κάνατε γι' αυτό. Και τρίτο ερώτημα. Για τις διαφορές ανάμεσα στις εργαστηριακές δοκιμές και στις πραγματικές ε, εκπομπές. Ποιος σας είπε να αναλύσετε αυτές τις διαφορές. Τι σας έκανε να αναλύσετε αυτές τις διαφορές. Πότε, επίσης, υπό ποιο επίτροπο έγινε αυτή η προσπάθεια. Πότε έγιναν γνωστές δηλαδή αυτές οι διαφορές. Εμείς ξέραμε ότι υπήρχαν αυτές οι διαφορές, όπως αναφέρατε και στο CARS 2020. Uh, όπως είπα νωρίτερα, κίνητρο των δύο μελετών που κάναμε ε, ε, ε, ήταν δύο διαφορετικά βασικά τα, κίνητρα. Το πρώτο ήταν ζητή, μας ζητήθηκε για να ελέγξουμε την τεχνική εφικτότητα των, του ελέγχου των ε, εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες των οχημάτων και το κίνητρο για την μελέτη που έγινε το 2013 ήταν να ελέγξουμε δύο μεθοδολογίες που είχαν προταθεί ως υποψήφιες. Πρώτον τα PEMS το άλλο ήταν οι δοκιμές ε, τυχαίου κύκλου. Um, ε, επαναλαμβάνω, αν ε, δείτε τα αποτελέσματα των δύο εκθέσεων, αν δείτε την, την σύνοψη και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αυτών, πουθενά δεν λέμε ότι υποπτευόμασταν τη χρήση συσκευών αλλίωσης στις μελέτες μας. Προσπαθήσαμε να ε, εξηγήσουμε για ποιο λόγο ενδεχομένως υπήρχαν αυτές οι ε, διαφορές και στόχος μας ήταν πάντοτε να ε, ενισχύσουμε την στιβαρότητα των ελέγχων σε πραγματικές συνθήκες. Εμείς δηλαδή είχαμε ως στόχο να βελτιώσουμε τις δοκιμές για να βελτιώσουμε ε, τις ε, διαδικασίες και να αποτρέψουμε τη χρήση συσκευών αλλίωσης. Ε, πουθενά όμως δεν λέμε ότι υποπτευόμασταν, είχαμε υποψίες ότι ενδεχομένως οι διαφορές αυτές να οφείλονταν στη χρήση συσκευών αλλίωσης. Μπορείτε να μας πείτε όμως πότε και ποιος ε, σας έδωσε αυτό το κίνητρο. Ε, Εντολή για την πρώτη μελέτη μας δόθηκε από την Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ 2004 με 2007 και τα αποτελέσματα ε, στα οποία καταλήγαμε τα συζητούσαμε πάντοτε με τις υπηρεσίες όχι μόνο με την ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων αλλά και με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ε, επίσης αυτοί χρηματοδότησαν ε, τις μελέτες οπότε ε, τους ενδιέφεραν τα αποτελέσματα και ήμασταν σε διαρκή επαφή μαζί τους γιατί στην πραγματικότητα είχαν συμμετάσχει ενεργά και εκείνοι στην ανάπτυξη του ερευνητικού προγράμματος. Είχαμε δηλαδή μια συνεχή επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορώ να σας δώσω δηλαδή μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωραία. Πάμε στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Κύριε Σκάρενς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μία λέξη έχω να πω. Wow. Διαβάζω και βλέπω τι κάνετε. Το 2004 είπατε ότι ξεκινήσατε αυτές τις πραγματικές μετρήσεις και το 2007 διαπιστώσατε ότι ε, υπήρχαν ε, αυτές οι διαφορές κατά 4 έως 7 φορές. Εντυπωσιακό. Ε, έχουμε αυτήν την ε, κλιματική πολιτική που μας λέει ότι πρέπει να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και ταυτοχρόνως συνειδητοποιείτε εσείς ότι ενώ προσπαθούμε να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα ξαφνικά τα οξύδια του αζότου απογειώνονται και σας πήρε δύο χρόνια, μέχρι το 2012, ε, μια μελέτη δημοσίευσα το 2011, ε, πραγματικά, αν ε, οι πολιτικοί σας έλεγαν μην το βγάλετε στη δημοσιότητα, αν οι αυτοκυβερνητικοί σας έλεγαν το ίδιο, ή μήπω τελικά απλά είχαμε ένα πλήρως αναποτελεσματικό σύστημα, όπου παρά το γεγονός ότι έχουμε επιστημονικά δεδομένα, εσείς ε, δεν ε, καταλήγετε στα συμπεράσματα που, που έπρεπε, γιατί εσείς ελέγχατε και ξαναελέγχατε και σας πήρε χρόνια όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε οι πολιτικοί λένε, οι αυτοκινητομηχανίες σας λένε μην μη το δημοσιεύσετε αυτά, ε, αυτός ήταν ο, ο λόγος ή απλά το σύστημα που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν απλά πάρα πολύ αργοκίνητο και αναποτελεσματικό. Όχι, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά που κάναμε και αυτά στα οποία καταλήξαμε ήταν ε, ε, μία από τις πιο προηγμένες στον κόσμο δοκιμές. Και πρέπει να αναγνωρίσετε ότι όταν ξεκινήσαμε με τα PEMS για τα βαρέα οχήματα, ξεκινήσαμε με εξοπλισμό που είχε βάρος έως και 100 κιλά και Μάλιστα χρειάστηκαν 78 χρόνια ερευνών για να φτάσουμε σε αυτό. 7 έως 8 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό και ε, καταλήξαμε σε νομοθεσία το, το 2007, τον 615, με τον, τον κανονισμό αυτόν η Κομισιόν ε, έδωσε τη δυνατότητα βελτίωσης και ενίσχυσης των δοκιμών. Έπρεπε λοιπόν να πάρουμε υπόψη μας τι υπήρχε ε, και λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγές μας και τι κάναμε τελικά. Κοιτούσαμε, είδαμε ότι αυτά που είχαμε ήταν ήδη κάποιες επιτυχίες και προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε αυτό που είχαμε στα ελαφρά οχήματα εξετάζοντας και διάφορους άλλους παράγοντες. Άρα, αν δείτε όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, ο χρόνος που μας πήρε να προσαρμόσουμε τα PEMS από τα βαρέα οχήματα στα ελαφρά οχήματα ε, ήταν περίπου 4,5 χρόνια. Ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι έγιναν και συνεδριάσεις στην Κομισιόν τεχνικών ομάδων, η ομάδα εργασίας RD, RDLDV, τα άλλα τρία χρόνια ε, τα αφιερώσαμε στην έρευνα για την προσαρμογή του ΠΕΜΣ και την επιλογή μεταξύ αυτών των τεσσάρων μεθόδων ε, για τις μετρήσεις ΠΕΜΣ. Έπρεπε να γίνουν συζητήσεις ε, και στη συνέχεια έπρεπε να γίνουν και δοκιμές. Όλα αυτά λοιπόν μαζί ε, πήραν όλο αυτόν τον χρόνο. Άρα δεν σας είπε η αυτοκίνητο βιομηχανία ή η πολιτική. Απλά το κάνατε όλο αυτό για να φτάσετε σε βάσιμα επιστημονικά συμπεράσματα. Άρα εσείς λέτε ότι εμείς οι πολιτικοί βιαστήκαμε να ε, καταπολεμήσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα χωρίς να ε, περιμένουμε να δούμε τι αντίκτυπο θα είχε μια τέτοια επιλογή ε, στις, στις άλλες ε, χημικές ονόσεις, για παράδειγμα στα οξύδια του αζότου. Αυτό λέτε. Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι βελτιωθήκαμε και μειώσαμε το χρόνο και ε, ε, μέσα σε πέντε χρόνια καταφέραμε και κάναμε αυτή την προσαρμογή και έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία πλέον στο πλαίσιο των δοκιμών εκπομπών και έτσι δεν χρειαζόμαστε πλέον τόσο πολύ χρόνο ακριβώς γιατί έχουμε πείρα πλέον. Thank you, uh, Κύριος Ευχαριστούμε πολύ την, ε, ε, την κυρία Αλκουντέρη για τις γραπτές της απαντήσεις. Μας βοήθησαν πολύ. Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των διατάξεων παράκαμψης, ε, Κάνετε μια διάκριση ανάμεσα στα ελαφρά και τα βαρέα οχήματα και αναφέρετε στο έγγραφό σας ότι χρησιμοποίησατε ε, επαγωγική λογική που βασίζεται στην εμπειρία σας και στην ιστορική ανάλυση των... της εφαρμογής του κανονισμού του 2007. Όμως το 1998 οι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη είχε βάλει πρόστιμο σε αυτοκινητοβιομηχανίες για τέτοιου συσκευέ σε βαρέα οχήματα και το 2004 βέβαια. βέβαια, ε, όταν χρησιμοποιούσαμε, χρησιμοποιούσατε τα PEM σε βαρέα οχήματα, είδατε σε τι οφειλόντουσαν οι διαφορές. Ε, γιατί δεν συνδέθηκαν τα όσα συνέβαιναν στο, στα βαρέα οχήματα με αυτά με τις διαφορές που βρίσκεται στα ελαφρά οχήματα. Καταλαβαίνω ότι η τεχνολογία θα έπρεπε να προσαρμοστεί, αλλά η εμπειρία με τα βαρέα δεν θα έπρεπε να μας διδάξει και για τα ελαφρά οχήματα. Uh, uh, Χρησιμοποιήσαμε την ε, εμπειρία μας με τα πέμψη στα βαρέα οχήματα ε, όταν ξεκινήσαμε τη δουλειά μας στα ελαφρά οχήματα. Αλλά θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στο συνάδελφό μου για να σας εξηγήσει πώς περάσαμε από το ένα στο άλλο. Not in extent, just very ε, εν συντομία όμως παρακαλώ, έτσι. Μην επεκταθείτε ιδιαίτερα. Καταρχήν, αυτό που κάναμε στα βαρέα οχήματα δεν ήταν μια μεθοδολογία, ήταν δοκιμές, δεν ήταν μεθοδολογία για τον εντοπισμό τέτοιων διατάξεων παράκαμψης. Ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα, έτσι. Χρησιμοποίησαμε τον ίδιο εξοπλισμό και παρόμοιες μεθοδολογίες για τα επιφατικά οχήματα. Καταρχήν, για κάποιες βασικές ιδέες που είχαμε στο πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος, ε, για οχήματα που κυκλοφορούν στις πόλεις και μετά τις πρώτες δοκιμές αντιληφθήκαμε ότι το πρόβλημα που έχουμε με το αοξίδιο του αζότου δεν το βρίσκουμε με άλλους ρήπους ε, και, και δεν το έχουμε και τόσο πολύ με τα βενζινοκίνητα οχήματα. Συζητήσαμε λοιπόν με την Κομισιόν τις Γενικές ε, περιβάλλοντο και Επιχειρήσεων και αρχίσαμε να αναπτύσσουμε τη μεθοδολογία. Ε, σαφές, σαφές ότι η μεθοδολογία για τα βαρέα επηρεάσει τη μεθοδολογία στα ελαφρά. Γιατί όμως δεν χρησιμοποίησατε και την παγωγική σα λογική έτσι ώστε να συμπεράνετε ότι δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είχαν βρει τέτοιου διατάξει από το 1998 και είχαν επιβάλει πρόστιμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και για τα ελαφρά οχήματα. Κανείς δεν συζήτησε, δεν έθεσε το θέμα της ύπαρξης τέτοιων διατάξεων σε ελαφρά οχήματα. Όχι, είναι η απάντηση της κυρίας Κουντέρη. Το θέμα είχε τεθεί στο τέλος δεκαετίας του 90, όπως είπατε. Αλλά ε, υπήρχαν απόλυτα λογικές εξηγήσει σε σχέση με τις δοκιμές εντοπισμού διατάξεων παράκαμψης. Γνωρίζαμε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς ε, ε, εντοπίζουμε μόνο συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένους τύπους συνθήκων οδήγησης. Οπότε χρησιμοποιούσαμε τις ΠΕΜΣ για να βελτιώσουμε το σύστημά μας, τη μεθοδολογία μας. Και επιβεβαιώσαμε ότι δεν αρκούν τα εργαστηρια... οι δοκιμές. Ωραία, αλλά και πάλι δεν απάντησατε την ερώτησή μου. Δεδομένου ότι οι Πολιτείε έβαλαν πρόστιμο για αυτό είναι ακριβώ ακριβώ το πρόβλημα ε, στους, κατασκευαστές εκεί στις ΗΠΑ. Ε, αυτό δεν θα ήταν αρκετό να σας οδηγήσει στο να σκεφτείτε ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει και εδώ και στα ελαφρά οχήματα. Δεν σας πήρε τόσα χρόνια. Ναι, η νομοθεσία μας ε, ε, δεν προβλέπει η Κομισιό να κάνει τον αστυνόμο. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα αυτή, έχουν τις τεχνικές αρχές μέσω των οποίων γίνεται αυτός ο έλεγχος και η εφαρμογή του νόμου. Οι εθνικές αρχές πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση και να επιβάλλουν πρόστιμα ενδεχομένως. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν το 2007 και τώρα με την αναθεώρηση του πλαισίου τύπου έγκρισης, έγκρισης τύπου, συγγνώμη, παίρνει σιγά σιγά περισσότερες αρμοδιότητες έτσι ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ε, χρειάστηκε να υποβάλουμε και επαρκείς αποδείξεις έτσι, για να ε, γίνει αυτή η μεταφορά αρμοδιότητας, η εκχώρηση. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που απαντάτε στα ερωτήματά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντοτε να διακρίνουμε μεταξύ ερωτημάτων που αφορούν την διαφορά μεταξύ των ε, ε, εργαστηριακών και των πραγματικών εκπομπών και σε ερωτήματα που σχετίζονται με αυτές τις συσκευές αλλίωσης. Και θέλω να επανέλθω σε αυτό το λογισμικό αλλήλωση. Μόλι υπόθηκε από συνάδελφο ότι από το 1998 οι αμερικανικέ αρχέ είχαν επιβάλει πρόστιμα σε αυτοκινητοβιομηχανίες για, ε, για τη χρήση τέτοιου είδου λογισμικού και μάλιστα τα πρόστιμα αυτά ε, ήταν εν μέρη και πολύ βαριά. Ε, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξή. Αυτό πρέπει να είχε σκάσει εδώ στην Ευρώπη σαν ε, βόμβα. Ε, ποιος, τι θα εμπόδιζε τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να χρησιμοποιήσουν ε, παρόμοιες ε, συσκευές ή διατάξεις. Ε, αυτές, αυτές οι, αυτά τα νέα για το τι συνέβαινε στην Αμερική δεν μπορεί να μην, ε, να μην έφτασαν στα αυτιά σας κάποια στιγμή. Οπότε ε, ε, ξαναθέτω και εγώ το ερώτημα. Ποτέ δεν μπήκατε στη διαδικασία να σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία εσωτερικά στο κοινό κέντρο έρευνας για το τι γίνεται. Υπενθυμίσω ότι ο ρόλος μας είναι να δώσουμε επιστημονικά στοιχεία. Κάνουμε έρευνα κατόπιν εντολής που μας δίδεται. Και να υπενθυμίσω ότι εκείνη την εποχή η Κομισιόν δεν είχε τέτοιο αστυνομευτικό ρόλο και ούτε έχει ακόμα. Γινόταν πάντα έρευνα, μα πάντα για να πετύχουμε κάτι σε επίπεδο πρόληψης. Δεν θεωρούσαμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το γιατί υπήρχαν διαφορές ανάμεσα αυτά που μετράμε στο εργαστήριο και στις ε, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Κάναμε πάντα έρευνα προκειμένου να βελτιώσουμε τις εκπομπές, το, τις δοκιμές εκπομπών, ούτω ώστε να μειωθούν τελικά οι εκπομπές των οχημάτων. Αυτή την εντολή είχαμε ανέκαθεν. Ναι, αλλά ισχυρίζεστε ότι είστε ερευνητικό κέντρο. Εγώ ήμουν κάποτε υπεύθυνο για 86 ερευνητικά κέντρα και οι διευθυντές αυτών των ερευνητικών κέντρων που γνώρισα εγώ ε, θυμάμαι ότι είχαν μια φυσική περιέργεια και δεν μου είπαν ποτέ ότι, εγώ, ότι εμείς ερευνούμε μόνο πράγματα που, για τα οποία έχουμε πάρει εντολή. Οπότε εγώ αναρωτιέμαι, είστε πραγματικά ερευνητικό κέντρο ή είστε σε τελική ανάλυση ε, ένα τμήμα, μια υποϋπηρεσία ενός ε, ανώνυμου μηχανισμού ε, Uh, Όχι, είμαστε το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Κάνουμε έρευνα για να βοηθήσουμε την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικές και να την εφαρμόσει την πολιτική της και να αξιολογήσει την εφαρμογή της πολιτικής. Αν κοιτάξετε την έρευνα που έχουμε κάνει, αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ε, κάποια νομοθετικά πλαίσια. Ήδη το 2007 αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια πρόληψης της δημιουργίας τέτοιων συσκευών αλλίωσης και ο ρόλος μας ήταν να βοηθήσουμε ούτω ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς το νομοθετικό πακέτο για την πρόληψη στα πλαίσια της εντολής που έχουμε. Με την εργαστηριακή μας προσπάθειες, με την μεθοδολογία για σενάρια εργαστηριακών δοκιμών, με την ανάλυση των ε, εκπομπών μέσω του συστήματος PEPS, του φορητού αυτού συστήματος ελέγχου εκπομπών, πάντα στα πλαίσια της ανεξαρτησίας μας και γι' αυτό τα αποτελέσματά μας είναι πάντα δημόσια, διαφανή Τώρα, από το 2011 και το 2013 είχαμε αποτελέσματα, ε, και τα βλέπαν όλοι. Ε, και εμείς και η Κομισιόν και οι υπόλοιποι, οι πάντες. Υπήρχαν διαφορές, αλλά που δεν ήμασταν σίγουροι ότι οφείλονταν και δεν οφείλονται. Θα Χρειαζόταν δεν και καλά να οφείλονται σε τέτοιες συσκευές αλλίωσης. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ε, δεν είναι δική μας ευθύνη και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο δεν έχουμε την εξουσία και την αρμοδιότητα να εφαρμόσουμε οτιδήποτε. Έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία είναι διαφανή, είναι στη διάθεση όλων κτλ. Δουλεύουμε με βάση μία εντολή. Ευχαριστώ. Όσο και περισσότερο ακούμε, τόσο περισσότερες ερωτήσεις ε, προκύπτουν. Ε, αν υποψιαζόμαστε κάτι. Τι πρωτόκολλο έχετε. Τι κάνετε δηλαδή συστηματικά όταν υπάρχει ας πούμε, κάποια ανομαλία, υποψία ανομαλία, στα λοιπά, δεν έχετε κάτι που να προβλέπετε στο πρωτοκόλλο σας. Για την, στην απάντηση στην ερώτηση 5α ε, λέτε ότι έγιναν, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές δοκιμές για να διαπιστωθούν οι ανομαλίες και πρέπει να δούμε αν υπάρχει ε, παράτυπη, παράνομη ας πούμε εφαρμογή και χρήση τέτοιων συσκευών αλλίωσης. Δηλαδή, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης ας πούμε των συσκευών αυτών όπως προβλέπει το άρθρο 5.2 του Κονισμού. Και τι χρειάζεται κάποιος ε, να κάνει ούτως ώστε να τροποποιηθεί το σημείο αυτό για να συμμορφούνται με τις προϋποθέσεις. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας ορισμός στον κανονισμό για το τι είναι η ε, διατάξη παράκαμψης και υπάρχει και μια μισή πρόταση στον κανονισμό υπό ποιε προϋποθέσεις ενδέχεται να επιτρέπονται αυτές οι συσκευές αλίεσης. Δεν έχουμε κριτήρια αξιολόγησης στον κανονισμό αυτή τη στιγμή και επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση των αυτοκινητοβιομηχανών να δώσουν στις αρχές ή στην Κομισιόν πληροφορίες για το ποια ε, τι είδους συσκευές αλλίωσης έχουν εγκαταστήσει και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται. Άρα αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κανονισμό, αλλά βρίσκονται υπό επεξεργασία για να ενσωματωθούν στον κανονισμό. Ε, υπάρχει κάτι άλλο επιπλέον που πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε νομοθετικά για να βεβαιωθούμε ότι θα καλύπτονται όλοι οι τομείς ε, ε, για να αναλαμβάνονται οι απαραίτητες δράσεις σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ανομαλιών. Υπάρχει μια πρόταση για ένα νέο ε, πλαίσιο έγκρισης τύπου το οποίο θα προβλέπει και επιτήρηση της αγοράς και χρήση σε πραγματικές συνθήκες από την Κομισιόν. Θα διενεργούνται δηλαδή δοκιμές όταν θα διατίθενται προϊόντα στην αγορά. Ένας μηχανισμός δηλαδή που θα επιτρέπει στην Κομισιόν να κάνει δικούς, δικές της δοκιμές που αυτή τη στιγμή επί του παρόντος δεν βρίσκονται, δεν εμπίπτουν στην εντολή της Κομισιόν αλλά στην εντολή της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Με αυτές τις δοκιμές ε, είμαστε σχετικά σίγουροι ότι το νέο βελτιωμένο πλαίσιο έγκρισης τύπου θα, ε, στις, ε, στα κράτη-μέλη θα ε, αποτελεί έναν πρόσθετο μηχανισμό ελέγχου που θα μας δίνει τη δυνατότητα αν κάποια συσκευή αλλίωσης δεν εντοπιστεί από ε, κάποια δοκιμή, να εντοπιστεί σε δεύτερο στάδιο στον ε, μηχανισμό ελέγχου που έχουμε ε, προτείνει. Η κυρία Κλειούνεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε το Κοινό Κέντρο Έρευνας που είναι εδώ μαζί μας. Η Κομισιόν ε, μας ανέφερε ότι είχε αυτό το μηχανισμό ελέγχου με βάση τα, τα και διαπιστώσαμε, συνειδητοποίησαμε ότι δεν επαρκεί τελικά αυτό. Ε, θα μπορούσαμε να σας ζητήσουμε την... Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να ζητήσουμε βοήθεια από εταιρείε που ε, διαθέτουν ε, τέτοιον φορητό εξοπλισμό για την δοκιμή εκπομπών ελαφρών οχημάτων. Υπάρχουν δεχομένως πολιτικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Και επίσης κάτι για τις δοκιμές σας. Δοκιμές σας. Στην, στις μετρήσεις εκπομπών οξυδίων του ε, αζότου σας ε, ποιες είναι, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες αβεβαιότητας που σχετίζουν, συσχετίζουν, που, που μάλλον σχετίζονται με, το, τα PEMS. Αναπτύσσεται κάποιο σύστημα για τη μείωση των αβεβαιωτήτων των μετρήσεων. Είπατε ναι, πώς ακριβώς το κάνετε και ε, ποιο είναι το τρέχον ε, ποσοστό αβεβαιότητας για τις μετρήσεις οξυδίων του αζότου. Και μια μικρή άλλη ερώτηση γιατί πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν έγκριση για την ευρωπαϊκή αγορά στο Λουξεμβούργο, παρότι καμία από αυτές τις αυτοβιομηχανίες δεν έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή. Η αβεβαιότητα είναι γύρω στο 20-30%. Ο άλλο ίσως θα μπορούσε να μα εξηγήσει γιατί υφίσταται τέτοια αβεβαιότητα και τι έρευνα κάνουμε για να μειωθεί αυτό το ποσοστό. Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές ανάμεσα σε δοκιμές στο εργαστήριο και σε πραγματικές συνθήκες. Ε, το, οι δοκιμές διαρκούν, είναι ενό κύκλου στο εργαστήριο και διαρκούν 20 λεπτά. Ε, οπότε ε, ε, ε, εκεί είναι δυνατόν να, διατηρούν; να έχουμε μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις συσκευές μας. στο δρόμο χρειαζόμαστε ε, μάλλον χάνουμε την ακρίβεια των ε, οργάνων μας, ε, δηλαδή το μηδέν μετακινείται επειδή το όχημα μετακινείται και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως, να είμαστε πλήρως 100% ακριβείς στις μετρήσεις μας στο δρόμο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή την αβεβαιότητα. Το 20-30% είναι μέγιστο, έτσι, δεν σημαίνει ούτε ότι είναι μεσοσόρος, ότι είναι μόνιμο. Τώρα, γιατί στο Λουξεμβούργο. Δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματος των βιομηχανών γιατί χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο. Υπάρχει επιστημονικός λόγος. Όχι. Είναι η απάντηση. Και ο Όχι. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τα οξύδια του αζότου. Ποια είναι η απάντηση. Ε, στις μετρήσεις σας για τα οξύδια του αζότου, ε, ποια είναι η αβεβαιότητα για τα, με με τις φορητές συσκευέ μετρήσεων. Και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να μειώσουμε αυτά τα ποσοστά βεβαιότητας. Ε, Σα είπα ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη χρήση συσκευών μέτρηση στο εργαστήριο σε στάσιμες ε, συνθήκες στασιμότητα και σε, ε, αφενός και αφετέρου σε ένα αυτοκίνητο που κινείται και σε διαφορετικό περιβάλλον. Ε, η αβεβαιότητα οφείλεται στην μετακίνηση του ουδέτερου σημείου των συσκευών μέτρησης στην απώλεια των ρυθμίσεων δηλαδή. Συζητήσαμε με ε, κατασκευαστές για να δούμε αν μπορούν να βελτιωθούν αυτά τα όργανα. Ε, μιλώ για κατασκευαστές ε, εξοπλισμού, έτσι, όχι αυτοκινήτων, και μας είπαν ότι ναι, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις συσκευές μέτρησης, τις φορητές μέτρησης. Τούρμες. έδωσα ένα έγγραφο για να καταλάβω την ερώτησή μου. Ε, κύριε Κουντέρη, ε, είναι σωστό να πω ότι η, η Γενική Διεύθυνση ε, Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η αρμόδια και η δική σας διεύθυνση F είναι αρμόδια για αυτή την έρευνα για τα φορητές ε, συσκευές μέτρησης. Οπότε εσείς η ίδια για 15 χρόνια ήσασταν στη Γενική Διεύθυνση G, έτσι. Το, το Νοέμβρη ε, διοριστήκατε διευθύντρια στην Α. Οπότε από, από αυτή την πλευρά δεν είχατε άμεση ε, συμμετοχή ούτε και πληροφορίες από πρώτο χέρι, έτσι δεν είναι για όλα όσα συζητούμε. Δηλαδή εσείς προσωπικά ε, ποτέ δεν συμμετείχατε σε καμία συνάντηση σχετική, έτσι δεν είναι. Πρόεδρος, κύριε Τούρμες, Ε, προσκαλούμε συγκεκριμένους ανθρώπους ε, και αν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι έρχεται κάποιος άλλος ο, όταν ποιος, ποιος σας ζήτησε, να εκπροσωπήσετε το JRC εδώ σήμερα. Να σας εξηγήσω το ρόλο μου καταρχήν. Είμαι γενική, ε, είμαι διευθύντρια ε, για το συντονισμό ε, πολιτικών. Οπότε χρειάζεται να εντοπίζω θέματα τα οποία, στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε και να αναπτύσσω ένα πρόγραμμα εργασίας για να βοηθήσουμε την Κομισιόν. Οπότε εγώ πρέπει να καταλαβαίνω πολύ καλά όλα όσα συμβαίνουν στο JRC. Ναι, πράγματι, ήμουν αλλού και ασχολιόμουν με άλλες πτυχές. Ε, οι σπουδές μου ε, είναι σχετικές, είμαι μηχανικός, καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα και παρακολουθώ το θέμα αυτό από τότε που μου ανακοίνωσαν ότι θα διοριστώ. Όχι πριν από δύο μήνες. Από πέρσι είμαι διευθύντρια. Από τον Νοέμβριο. <laughs> Και ε, μου ανακοινώθηκε ότι θα διοριστώ το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν παρακολουθώ το ζήτημα αυτό πολύ στενά. Και το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ε, ήταν να ανακοινώσω πληροφορίες ε, για τις ε, δύο έρευνες που είχαμε, γιατί μας το ζητούσαν πολύ. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν <laughs> να ασχοληθώ με αυτά τα αιτήματα πληροφόρηση σε σχέση με τις δύο μας μελέτες. μετά τα όσα τα δυσάρεστα που έλαβαν χώρα, ε, αλλάξαμε την ημερομηνία της συνεδρίασής μας, ε, για, ενώ της σημερινής σας συνεδρίασης, ε, ο, ε, οπότε δεν, δεν μπόρεσε να είναι παρόν ο Γενικός Διευθυντής. όταν ορίστηκε η σημερινή ημερομηνία πλέον δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ, είχε μια άλλη συνάντηση και γι' αυτό το λόγο μου ζήτησε ο Γενικός Διευθυντής μου να έρθω εγώ. Ε, διότι ε, εγώ είμαι υπεύθυνη για τον συντονισμό στήριξης των πολιτικών. Ο κ. Γκάσεμπερκ με ε, συνοδεύει όμως που είναι επικεφαλής του τμήματος, τμήματάρχης δηλαδή, στο τμήμα το οποίο ασχολήθηκε με τις δοκιμές αυτές και με την έρευνα. Προκειμένου να με βοηθήσει να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ποιος ήταν διευθυντής ενέργειας και μεταφορών τα τελευταία χρόνια. Ο Τζοβάνι Ντισάντι και είναι ακόμα διευθυντής. Είστε σίγουροι ότι είναι ακόμα διευθυντής. Εξ όσων γνωρίζω μέχρι σήμερα είναι. Γιατί η δική μου πληροφορία είναι ότι ο κ. Ντισάντι μετακινήθηκε πριν από μερικές ημέρες. και μου αναφέρουν ο κ. Ντεσάντη ήταν διαθέσιμος για τη συνεδρίαση αυτή σήμερα και ότι ο κ. Σούτσα ε, επέλεξε να μην στείλει έναν εδώ σε εμά, έναν από τους ανθρώπους που πιο πολύ κατανοούν το θέμα. Σκοπίμως. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά ειλικρινά δεν περιμένω ότι θα πάρω ακριβείς απαντήσεις από κάποιον που δεν έχει ε, εμπειρία από πρώτο χέρι. Γιατί εμείς θέλουμε να δούμε ποιες ήταν οι αδυναμίες από τους ανθρώπους που ήταν παρόντες. Είναι αλήθεια ότι το, τα PEMS που χρησιμοποιήθηκαν από τις Αμερικανικές αρχές ε, αναπτύχθηκαν εν μέρη από το GRC. Είναι αλήθεια ότι ο ICCT, ότι το προσωπικό του ICCT δούλεψε στο GRC κάποιες, σε κάποιες περιόδους στο παρελθόν και κατά κάποιο τρόπο απομακρύνθηκε από εκεί. Και όταν λέτε ότι δεν υπήρχε ποτέ κανένας είδους ε, αποδεικτικό στοιχείο και κανένας δεν υποπτέθηκε στο GRC ότι είναι υπάρξει τέτοιων συσκευών εξαπάτησης, να σας διαβάσω από τη δική σας έκθεση του 2013 που λέει ε, οι δοκιμές Κύριε Τούρμε, λέει πρόεδρος, κύριε Τουρμέ, δεν, έχετε χρόνο για, δεν έχουμε χρόνο για απάντηση. Αφήστε το για την, τον επόμενο γύρο. Μία, μία, μία φράση θέλω να διαβάσω. Και μετά θα δούμε πόσο, χρόνο, πόσο χρόνος μένει. Δυστυχώς μιλούν ο ένας πάνω στον άλλο μιλητές. Οι συσκευές PEMS θα είναι πιο αποτελεσματικές στην πρόληψη και ε, της χρήσεως ε, στρατηγικών εξαπάτησης. Το 2013 λοιπόν ε, ο, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, του κλείνει το μικρόφωνο. Κύριε Εύη, οπότε, ο κ. Στουρμες, οπότε το GRC υποπτευόταν την ύπαρξη τέτοιων στρατηγικών ε, παράκαμψης. Κύριε Εύη. Να πάρω εγώ τον λόγο τώρα. Θα μιλήσω Ιταλικά. με βάση τα όσα μας απαντήσετε, 6β, οι τεχνολογίες που μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές οξυδίων του αζότου σε πραγματικές συνθήκες ε, εκπομπών με βάση τα όρια του καονισμού του 2007. Αυτά τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ήδη στην αγορά. Στην 11β για την ακρίβεια των PEMS μπορούμε να μειώσουμε ε, την αβεβότητα στο 10-15%. Με βάση αυτά τα στοιχεία δεν νομείτε ότι η εισαγωγή ενός παράγοντα διόρθωσης που μιλάει για 168 ε, μικρογραμμάρια ε, μέχρι το 2020 δεν έχουν κανένα νόημα. Επίσης, αν έχω άλλο χρόνο, να ρωτήσω το εξής. Για τα, όρια εφαρμο... τα νόμιμα όρια εφαρμογών αυτό των συσκευών αλλίωση. Στην απάντηση 10. Μιλάτε για απουσία πραγματικών ορίων που μπορούν να δικαιολογούν την προσφυγή σε εξαιρέσεις. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που εμποδίζουν τους κατασκευαστές να που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να βάλουν νομίμως ε, τέτοιες συσκευές, μπερδεύοντας τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη μιλάω για τα στοιχεία και τα αρχεία που έχουμε για, την, για τα αυτοκίνητα Audi. Sorry for taking so long. Δυσκολεύτηκα να παρακολουθήσω την ερώτηση. Να ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα που αφορά τις συσκευέ αλλίωσης και τις ε, μεθοδολογίες για να τις εντοπίσουμε. Είναι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή. Γιατί πρέπει να έχουμε πρόσβαση όχι μόνο σε hardware, αλλά σε λογισμικό και στην ε, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου, που διαχειρίζεται την ε, συμπεριφορά του κινητήρα και του συστήματος ε, καθαρισμού των καυσαερίων. Και δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα. Εάν θέλετε λοιπόν πραγματικά να, να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει μια τέτοια συσκευή, και όχι κάποιε στρατηγικέ που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστή για να προστατεύσει ας πούμε, τον κινητήρα, τότε θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το λογισμικό. Αλλιώ δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τέτοιε συσκευέ στο αυτοκίνητο. Αλλιώ και έχουμε απλώ ενδείξει. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι σίγουρα υπάρχουν αυτέ οι συσκευέ. Και για τα επίπεδα αβεβαιότητα των PEMS, των φορητών συσκευών. Στο 11β σας διάβασα ότι μπορούμε να, μειώσουμε αυτό το επίπεδο αβεβαιότητας ε, και να το φτάσουμε στο 10-15%. Ναι, το έχω ξαναπεί αυτό. Απαντώντα σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ο μεγαλύτερο λόγο αυτού του σφάλματος, είναι να περάσουμε από το 30% ας πούμε ε, σφάλματος ή αβεβαιότητας στο 15-20% ε, με βάση τα όσα λένε οι κατασκευαστές των ε, φορητών συσκευών. Ο διορθωτικός παράγοντας, επομένως που θεσπίζουμε, είναι πολύ μεγάλος. Δεδομένων των ποσοστών αυτών σφαλμάτων που έχουμε σήμερα. Ο παράγοντας συμμόρφωσης δεν συμπεριλαμβάνει το σφάλμα του, της συσκευής δοκιμής, αλλά μόνο της διαδικασίας δοκιμής. Γιατί μπορεί να έχεις διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας και αυστηρότητας των δοκιμών που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και που απαντάτε στα ερωτήματά μας. Να επισημάνω το εξής. Αυτά που ε, ε οι απαντήσεις που δώσατε και εδώ αλλά και γραπτός δείχνουν ότι το 2006-2007 είχατε ήδη υποψία ότι ενδεχομένως να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει χρήση συσκευών αλλίωσης. Αυτό σε συνδυασμό με, το, με αυτά που αναφέρθηκαν για το σκάνδαλο το 1998 στην Αμερική και το γεγονός ότι εκπονήσατε το 2013 μελέτη όπου αναφέρεται ότι ε, διαπιστώθηκαν υψηλότερες εκπομπές οξυδίων του αζότου ε, αν, ανεξάρτητα από το αν ε, οφείλονταν αυτές ε, σε ανεπάρκειες των ελεγκτικών μηχανισμών. Το 2013, έχοντας πλέον αυτές τις τεχνικές γνώσεις, ε, έχουν ένα ερώτημα επικοινωνιακού χαρακτήρα ή άλλος ποια είναι ακριβώς η ιεραρχία στην υπηρεσία σας. Το JRC δεν θα έπρεπε ή δεν θα όφιλε να ερευνήσει το θέμα με δεδομένο και το σκάνδαλο που είχε γίνει στην Αμερική ή έστω να συζητήσει εσωτερικά ε, το όλο θέμα και να καταλήξει σε ένα πρόγραμμα δράσεων. Ωραία. Ε, για, μα, αυτόν τον λόγο, ε, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα εργασίας RDE-LDV. Και συστήθηκε η ομάδα αυτή ε, μόλις ε, διαπιστώσαμε τις διαφορές μεταξύ των ε, δοκιμών PEMS και των εργαστηριακών δοκιμών. Η Κομισιόν μάλιστα διοργάνωσε και ένα ειδικό εργαστήριο, workshop και στη συνέχεια συνέστησε αυτήν την ομάδα εργασίας. Και Πέραν αυτών όμως έγιναν μια σειρά από ε, συναντήσεις προκειμένου να καταρτιστούν οι απαιτήσει για τα PEMS, ε, όλα αυτά που ε, συζητούμε ακόμη δηλαδή. Γίνονται διαρκώς συζητήσεις, τα βήματα συζήτηση αυτές είναι, είναι ανοιχτά στα κράτη-μέλη, στις αρχές και εμείς συζητούμε πάντοτε τα ευρήματα και τα πορίσματά μας ανοιχτά, δημόσια και στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών των ομάδων εργασίας αλλά και υποομάδων ε, εργασίας ε, που, στις οποίες ανατέθηκε να ε, αναλυθούν οι μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των δεδομένων PEMS. Η συζήτηση αυτή λόγω και της σύστασης της ε, ομάδας εργασίας RDE-LDV e, ε, ήταν πάντοτε ανοιχτή μέσω και των δημοσιεύσεων. Όλα τα πράγματα συζητιόντουσαν πάντοτε ανοιχτά. Ε, ειδικά στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας των Και όπως είπα είχαμε και εκπροσώπους των κρατών μελών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, των αρμοδίων αρχών από τα κράτη-μέλη κτλ. κτλ. Συνάδελφοι, θα περάσουμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Τρία λεπτά για κάθε ερώτηση παρακαλώ. «45 δευτερόλεπτα καθένα και περάστε κατευθείαν στην ερώτηση. Κύριο Μπίλετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομο θα είμαι. Ε, έπειτα από ε, όσα έγιναν το 98 ε, στις ΕΠΑ, ε, εντάξει είπατε ότι δεν είπατε να απαντήσετε ή να αναλάβετε κάποια δράση. Παρ' όλα αυτά, 15 χρόνια μετά τα όσα έγιναν στις ΗΠΑ. Ε, ε, ε, υπήρχαν λοιπόν κάποιε ενδείξει για τι Αμερικανικέ Αρχέ. Είχατε κι εσεί ενδείξει τέτοια για τη χρήση συσκευών αλλίωση. Οι Αμερικανικέ Αρχέ όμω τελικά ανακάλυψαν τι ακριβώ είχε πάει λάθο. Επρόκειτο ε, ε, τις εντόπισαν αυτές τις συσκευές αλλίωσης ή ε, ομολόγησε για παράδειγμα στη δική μας περίπτωση η Volkswagen ότι είχε χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους συσκευές αλλίωσης. Προφανώς γνωρίζει κανείς ότι η ανακάλυψη αυτών των συσκευών αλλίωσης στις ΕΠΑ δεν έγινε μέσω του, του ε, EPA του Οργανισμού για την ε, ε, Προστασία του Περιβάλλοντος έγινε από μη κυβερνητική οργάνωση και έτσι καταλήξαμε σε ομολογία. Με άλλα λόγια, στη ΣΥΠΑ υπήρχε το πλαίσιο που έδωσε τη δυνατότητα να κατανοηθεί ε, ο τρόπος με τον οποίο ε, τα πράγματα εξελίχθηκαν. Ε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της είπα είναι υποχρεωμένες να ε, δημοσιεύουν ή να κοινοποιούν τις στρατηγικές τους για την μείωση των εκπομπών. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Προληπτικά και για να μην ξαναγίνουν αυτά που ε, έγιναν το τελευταίο διάστημα. Και Θέλουμε δηλαδή από εδώ και πέρα να έχουμε μια εκ των προτέρων κοινοποίηση από την αυτοκινητοβιομηχανία για το πώς θα ε, μειώνουν τις εκπομπές από εδώ και πέρα. Όπως είπα στη ΣΥΠΑ, δεν ήταν ο οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος αυτός που ε, εντόπισε ανείχνευσε το, όλο σκάνδαλο. Ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία εντόπισε το πρόβλημα και τελικά οδήγησε στις εξελίξεις της γνωστές. θα επιμείνω. Γιατί είπατε ότι το GRC δεν είχε ε, ε, καμία ιδέα για το ότι χρησιμοποιούνταν τέτοιες συσκευές αλλίωσης. Μεταξύ 98 και 13 υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση. Το 13 ωστόσο η Κομισιόν φαίνεται να ομολογεί ότι κάτι συμβαίνει και ότι κάτι μάλλον δεν πάει και πολύ καλά γιατί σε έγγραφο εργασία τη Κομισιόν με ημερομηνία 2013 σε ένα σημείο εκεί όπου γίνεται λόγος για τις αδυναμίες των δοκιμών συνομόρφωση, η Κομισιόν λέει ότι κάποια οχήματα φαίνεται ότι έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να συμμορφώνονται μόνο στην ε, υποσυνθήκες δοκιμών. Επίσης υπάρχει, ε, υπάρχουν ενδείξει ότι κάποιοι κατασκευαστέ προσπαθούν τεχνιέντο να βελτιώσουν τι μετρήσει τους. Άρα υπήρχαν αποδείξεις το 1998 ότι κάτι συνέβαινε, κάτι δεν πήγαινε και πολύ καλά. Ίσως δεν χρησιμοποιούνταν διατάξεις παράκαμψης ή αλλίωσης, αλλά αν όλα αυτά τα στοιχεία δεν σας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι γίνεται κάτι παράνομο ή ότι χρησιμοποιούνται συσκευέ αλλίωσης, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα σας οδηγούσε σε τελική ανάλυση. Βλέπω ότι ε, ε, προσπαθείτε να ε, τεκμηριώσετε τη θέση και τη στάση του JRC, ότι δεν υπήρχαν δηλαδή βάσιμες υποψίες. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι θα ήταν δηλαδή βάσιμες υποψίες ε, για σας. Και δεύτερο ερώτημα, πώς μπορείτε συνεχώς να βελτιώνεστε, γιατί αυτό λέτε ότι το κοινό κέντρο έρευνα θέλετε διαρκώς να, να βελτιώνετε. Πώς μπορείτε να βελτιώνεστε αν δεν αναγνωρίζετε καν τις αδυναμίες ή τις ανεπάρκειες που είναι αναμφίβολο ότι υπάρχουν. Σχεδόν δύο λεπτά ε, πήρατε κύριε Ντάρη, λέει η τις ανεπαρκειες που ειναι αναμφιβολο οτι υπαρχουν σχεδον δυο λεπτα ε πηρατε κυριε νταρι λεει η προεδρος <clears throat> Επαναρχόμαστε στις διατάξεις ε, παράκαμψης. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν ε, συσκευές που είναι νόμιμες και άλλες που είναι παράνομες. Αλλά δεν είναι σαφές τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Ποια χρήση είναι νόμιμη, ποια χρήση είναι παράνομη. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί και το έχουμε λάβει υπόψη στην καινούργια πρόταση. Στο μέλλον, αν αυτή η πρόταση ευοδοθεί, ελπίζουμε ότι οι αρχές θα έχουν πλέον πληροφορίες από τις αυτοκινητοβιομηχανίες για το τι είδους συσκευές, διατάξεις και συστήματα έχουν εγκαταστήσει οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με ποιο σκοπό και έτσι θα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν. Δηλαδή, θα έχουμε πλήρη γνώση του τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει ο κατασκευαστής. Ο κ. Γκίζεκε, είναι εντυπωσιακό που αφενός τα PEMS ε, ε, προβάλλονται ως λύση και αφετέρου μας ε, αναφέρεται ότι έχουν αβεβαιότητα 30% η ε, περιθώριο σφάλματος. Τελικά πόσο ασφαλή είναι τα PEMS. Σύμφωνα με το JRC, ε, σύμφωνα με τα στοιχεία του JRC, λέτε ότι η διαφορά είναι μέχρι 30% σήμερα. Κομισιόν μιλούσε για 13 με 15 μιλιγράμμ. Ε, τα δικά σας ευρήματα ποια είναι. 15 μιλιγράμμ είναι το, 15 ε, μιλιγράμμ είναι το μέγιστο που μετράτε ε, μάλλον το μέγιστο σφάλμα συγγνώμη, αν 15 μιλιγράμμ είναι το μέγιστο σφάλμα ε, είναι ικανοποιητικό αυτό δεν κατάλαβα. Πού, πού τα βγάλατε αυτά τα 15 μιλιγκράμμ. Πού προέκυψαν. Ε, ε, ο παράγοντας συμμόρφωσης λέει 15 μιλιγκράμμ. No, was not. Uh, I haven't proposed anything. Um, uh, we have only said. Εγώ δεν πρότεινα κάτι, τίποτε, τίποτε. Εγώ λέω ότι στην ανάλυση της, του σφάλματος των φορητών συστημάτων ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ε, η αβεβαιότητα είναι με 30% όχι 15 μιλιγκράμμ ούτε 30 μιλιγκράμμ. Η ερώτησή μου ε, ε αφορά το εξής. Ε, πόσο, επηρεάζει η θερμοκρασία στην ομιμότητα των συστημάτων παράκαμψης. Αυτά τα συστήματα αυτοεξουδετερώνονται πάνω από τους 10 βαθμούς, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από, για το ποιες θερμοκρασίες ανάβουν ή σβήνουν τα συστήματα αυτά της, των κατασκευαστών. Γιατί όχι. Sie sind ich der... την εντολή σας, τη δική σας εντολή, βλέπω ότι ε, είστε ε, Ινστιτούτο Έρευνας ε, επιστημονικής έρευνας και παρέχει τέτοιου είδου υπηρεσίες. Δεν θα έπρεπε να ξέρετε ότι ε, για παράδειγμα το Υπουργείο Μεταφορών τη της ε, έχει στοιχεία τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για αυτό το θέμα. Um, the question is... Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Οι αυτοκινητοβιομηχανοί δεν αναφέρουν σε εμάς ε, τις στρατηγικές ελέγχου τους. Δεν μας ενημερώνουν ούτε για το ποιες θερμοκρασίες ε, ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τα συστήματά τους. Επιπλέον, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε κανόνες είδους πληροφόρηση ε, που συλλέγεται από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή αρχή. Λέτε ότι τέτοιου είδους πληροφορίες είναι διαθέσιμες, αλλά δεν ξέρω αν είναι τότε δεν ερευνήσαμε σωστά, αλλά αμφιβάλλω για το κατά πόσον είναι δημόσιες αυτές τις πληροφορίες. Ε, ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά χρειάζονται τέτοιου είδου συστήματα ενεργοποίησης απενεργοποίησης. Απάντηση. Το συζητήσαμε το θέμα ε, των τεχνολογιών ενεργοποίησης απενεργοποίησης. Ε, καταρχήν, στον τομέα των ε, κινητήρων ε, ε, οχημάτων εκτός δρόμου και στα βαρέα οχήματα. Υπάρχουν δυσκολίες με τις χαμηλές θερμοκρασίες, με τη χρήση καταλυτών. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ο καταλύτης δεν λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε ε, ενεργοποιείται μόνο σε ψηλές σχετικά θερμοκρασίες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες ο καταλήτης δεν λειτουργεί. Ε, με την έγχυση ουρίας ε, μπορεί να τον καταστρέψεις. Αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο σε χαμηλές θερμοκρασίες το σύστημα ε, δεν πρέπει να, να μετρά τις εκπομπές ακόμα. Ο... Μόνο όταν ο καταλήτης φτάσει στην θερμοκρασία ε, λειτουργίας του, τότε πρέπει να μετράμε τα οξύδια, γιατί αλλιώς είναι πολλά, πολύ ψηλά οι μετρήσεις μας. Με δύο λόγια, εσείς λέτε ότι χρειάζεται να υπάρχουν διάφορα παράρθυρα θερμοκρασιών, δηλαδή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς λειτουργούν τα συστήματα επεξεργασίας των καυσίμων. Και είναι σαφές ότι αν η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο, δεν λειτουργούν. Ε, τα ερωτήσει που θέτουμε είναι πολύ σημαντικέ. Γιατί ε, το καινούριο σύστημα εγκριστή που θα σα δώσει περισσότερε αρμοδιότητε και βασιζόμαστε σε εσά να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Οπότε, σα ρωτήσω το εξή. Έχετε αρκετά κονδύλια για να φέρετε σε πέρα σε αυτό το καινούριο ρόλο σας, που θα είναι τεράστιος. Δεύτερον, ε, έχετε επαρκή δυνατότητα να διδαχθείτε από αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα έχετε την αναγωγική ικανότητα που χρειάζεται. Ε, επίσης, θα χρησιμοποιήσετε δικό σας προσωπικό ή υπεργολαβία με εξωτερικούς συνεργάτες. Τρίτον, πώς θα συνεργαστείτε με τις εθνικές αρχές, διότι δεν, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουν να ελέγχουν την αγορά επειδή θα νομίζουν ότι το κάνετε εσείς και δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων και δράσεων. We have, um... Έχουμε διάφορα εργαστήρια. Τα μέλη της Επιτροπής, ε, όταν ε, έρθουν τον Ιούλιο να μας επισκεφθούν, θα τα δείτε. Έχουμε μια πλειάδα εργαστηρίων που προτείνουμε για να μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε αυτές τις επιπλέον αρμοδιότητες. Επίσης, αν η πρόταση εγκριθεί, θα προσθεθούν άλλα δύο εργαστήρια στην παλέτα μας. Επίσης, θα αυξηθεί το προσωπικό μας. Δεν αποκλείεται επίσης υπό την καθοδήγησή μας ε, να αναθέσουμε και σε εξωτερικούς συνεργάτες ε, με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες όμως ε, κάποια τμήματα. Θα ξεκινήσουμε πάντως με τα εργαστήρια που έχουμε στη διάθεσή μας και θα επεκταθούμε. Θα εκτιμούμε ότι θα μας πάρει περίπου δύο χρόνια ούτως ώστε να ελέγξουμε ένα κάποιο δείγμα και όταν εντατικοποιήσουμε, ο άλλος θα μας πει το μέγεθος του δείγματος, αλλά θα αυξήσουμε το μέγεθος του δείγματός μας, ε, επιταχύνοντας προσπάθειες, αυξάνοντας προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι οι εθνικές αρχές θα αισθανθούν ότι τους υποκαθιστούμε. Γιατί εμείς θα, δοκιμα... θα ελέγχουμε την επιτυχία της διαδικασίας συμμόρφωσης, ε, δουλεύοντας πάνω σε δείγματα. Είτε απευθείας, ε, σε απευθεία συνεργασία με τις αρχές, είτε κάνοντας επιλογή ε, οχημάτων από την αγορά, είτε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των αρχών. Καταλαβαίνουμε εμείς από οχήματα. Και αν χρειαστεί να ξεπεράσουμε το δείγμα, τότε Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και εξωτερική ανάθεση. ανάθεση. Η δουλειά αυτή όμως θα γίνεται πάντα υπό την εποπτεία μας. Ε, ο συνάδελφος σας μιλήσει λίγο για το, δείγμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ. Για τις εκθέσεις. Τα φορητά μηχανήματα, οι φορητέ συσκευέ είναι πολύ βαριά και επηρεάζουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Επίσης, χρησιμοποίησατε ε, παλιά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα με διάφορα χιλιόμετρα, ας πούμε. Ε, ο αριθμός των χιλιόμετρων που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο επηρεάζει τις εκπομπές του. Πάντα για τις εκθέσεις. Στη σελίδα 4 της έκθεσης του 2011 λέτε ότι για, τα, για τους, το, το πρότυπο ε, Euro 6 υπάρχουν διατάξεις ε, ούτως ώστε να γίνονται σεβαστά τα όρια των εκπομπών κατά τη διάρκεια έγκρισης τύπου υπό κανονικές συνθήκες. Ε, επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν ε, μηχανισμοί ε, switch off. Γιατί αλλάξατε γνώμη και στη σελίδα 31 της έκθεσης του 2013 λέτε ότι οι εξαιρέσεις αφήνουν περιθώρια ερμηνείας στις απαντήσεις που δίνετε. Λέτε ότι ακόμη και καλύτερες δοκιμές ε, δεν μπορούν να ε, αποκλείσουν τη δυνατότητα ε, χρήσης ε, τέτοιων συσκευών ε, παράκαμψης. Τι γίνεται με την νομοθεσία, μήπως ανοίγουμε έτσι το παραθυράκι για να παρακάμπτουμε την νομοθεσία, να μην τη σεβόμαστε κτλ. Um, I from the uh, devices. Για τα PEMS. Φτιάχτηκαν για να γίνονται δοκιμές ε, σε φορτηγά, όπου υπάρχει πολλής χώρος και η κατανάλωση του κινητήρα δεν είναι πρόβλημα. Και σε αυτή την περίπτωση το βάρος των συσκευών αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όντως θα ήταν καλύτερο να είχαμε πιο ελαφρές συσκευές για τα επιβατικά οχήματα. Όταν ξεκινήσαμε τις δοκιμές δεν είχαμε επιλογή, μόνο αυτό το σύστημα είχαμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα μεγαλύτερα οχήματα, πιο βαριά οχήματα και προσπαθήσαμε να εγκαταστήσουμε όλα τα συστήματα στο αυτοκίνητο. αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, οι συσκευές αυτές έγιναν και πιο μικρές, ε, πιο ελαφριές, πιο εύκολες στο χειρισμό. Δεν χρειαζόταν, ας πούμε, να γίνει βαθμονόμηση κτλ. Και, και, να έχουμε αέρια ειδικά για τη βαθμονόμηση τα λοιπά Ήταν πιο απλές συσκευέ. Ε, μιλήσατε για διαφορετικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με διαφορετικά χιλιόμετρα και κατά πόσο επηρεάζουν τις εκπομπές. Φυσικά, σημα, φυσικά επηρεάζουν. Τα πιο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα φυσικά έχουμε υψηλότερε εκπομπές αλλά αποκλείεται. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή, εδώ δεν μπαίνει το πρόβλημα των συσκευών αλλίωσης. Δηλαδή, άλλο, συσκευέ αλλιώ και άλλο το πρόβλημα των χιλιόμετρων που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο. Κύριε Σορίνιο, καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Το 2013 το εργαστήριό σα. Ε, ε, λέει ότι παρόλο ότι οι Ευρωπαϊκέ προδιαφέρειες γίνονται όλο και πιο αυστηρές, ε, τα αποτελέσματα ε, στα εργαστήρια συμμορφώνονται αλλά όχι και τα αποτελέσματα στο, σε μετρή στο δρόμο. Οπότε αυτό ε, δίνει την ε, δυνατότητα, ε, την, δημιουργεί την υπόνοια ότι χρησιμοποιούνται συσκευές παραποίησης. Είχατε λοιπόν λόγους να είσαστε φιλίποπτοι είχατε πολύ συγκεκριμένους λόγους. Στην πραγματικότητα όμως ε, δεν ακολουθήσατε αυτή την οδό. Είναι σημαντικό εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν ε, ήσασταν δυσπιστοί έναν των αποτελεσμάτων που βλέπατε. Δεν το καταλαβαίνω. Είπατε ότι δεν ήταν ο αντικείμενο της μελέτης σας, ούτε είχατε μελέτη. Ναι, ωραία, δεν είχατε ε, εντολή, αλλά είχατε υποχρέωση ενημέρωση κομισιών. Την ενημερώσατε, ποιον ενημερώσατε. Και αν ναι, αν ε, ενημερώσατε, γιατί δεν σας διεύρυναν την εντολή. Δεν θα έπρεπε να ζητήσετε την επέκταση ε, την, ε, της εντολής σας δεδομένου των όσων γράφετε στην έκθεσή σας. Um, Επανέρχομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα. Αλόης εξήγησε γιατί θεωρήσαμε ότι ενδεχομένως υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ΠΕΜΣ και των ε, εργαστηριακών αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Φυσικά οι υπηρεσίες μας ήταν πάντοτε ενήμερες. Ε, αλλά και γι' αυτό το λόγο άλλωστε ε, διοργανώσαμε και αυτό το workshop για να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα του, της πρώτης μελέτης. Αυτό έγινε στο, στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου της Κομισιόν, στο οποίο συμμετείχαν και διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ο λόγος ε, είναι επίσης ε, για το γιατί θέλαμε να βελτιώσουμε τις δοκιμές ήταν και ε, γιατί τελικά συστήσαμε αυτήν την ομάδα εργασίας RDE-LDV ε, που ήταν όπως είπα ανοιχτή ε, σε κράτη-μέλη, σε αυτοκινητοβιομηχανίες, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και στο πλαίσιο των συναντήσεων της οποίας πάντοτε συζητούσαμε τα πορίσματα των μελετών μας με ανοιχτό τρόπο ακριβώς για να βελτιωθούμε. Και γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε υπάρχει και η δέσμη RDE και η νέα πρόταση για την ε, έγκριση τύπου. Και θεωρούμε ότι από εδώ και στο εξής ε, όλα αυτά θα δράσουν προληπτικά ως προς ε, την ε, στρατηγική δοκιμών, αλλά θα βελτιώσουν και τη μεθοδολογία ε, PEMS και έτσι μαζί με την έγκριση τύπου θα έχουμε στο μέλλον ένα πολύ καλύτερο οπλοστάσιο για να προλαμβάνονται τέτοιου είδους φαινόμενα αλλά και για να κατανοούμε καλύτερα το, τις ε, διαφορές μεταξύ των πραγματικών και των εργαστηριακών δοκιμών και προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε ε, τις ε, πραγματικές, ε, τα, τις πραγματικές μετρήσεις. Η πρόεδρος λέει να είμαστε πιο σύντομοι. Η κυρία Σαρανόβα, Σαραντζόβα, συγγνώμη. Χαράντζοβα, την διορθώνει η Ευρωβουλευτή. Ευχαριστώ. Ρόλος της Επιτροπής μας είναι να διερευνήσουμε τις διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα αν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσει που καθορίζονται από τον κανονισμό του 2007. Εκεί οι κύκλοι δοκιμών πρέπει να ελέγχονται από την Επιτροπή και να προσαρμόζονται αν δεν είναι αποτελεσματικοί και να ε, διασφαλίζεται ότι θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες. Οι μελέτες σας, οι εκθέσεις σας του 2011 και του 2013 κατέδειξαν σαφώς ότι οι δοκιμές δεν ήταν επαρκείς για τα ελαφρά οχήματα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε απαντήσεις για... και να μας πείτε ότι η Επιτροπή πράγματι ανταποκρίθηκε στις απαιτήσει που έθετε ο κανονισμός ή τελικά απέτυχε να το κάνει. Επίσης, ποια είναι η γνώμη σας ε, για το αν η Κομισιόν εισήγαγε τους νέους, τις νέες δοκιμές ε, έγκαιρα, όπως ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός του 2007. Διαδικαστικά νομίζω ότι η Κομισιόν έκανε ό,τι έπρεπε και γι' αυτόν τον λόγο ε, ζήτησαν οι υπηρεσίες της Κομισιόν αυτές τις δύο δοκιμές την ε, δημόσια ε, έκθεση του 2011 αφενός που η εντολή δόθηκε νωρίτερα βεβαίως και η οποία μελέτη ε, ζητήθηκε προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές μέσω της βελτίωσης της δοκιμής των εκπομπών. Για τις ε, δοκιμές κύκλου που αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε. Στη δέσμη RDE υπάρχει η ετήσια εντολή να αναθεωρούμε και αυτή τη διάσταση και αυτό λοιπόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από εδώ και πέρα στο, στους τέσσερις άξονες του RDE και το ίδιο ισχύει και για τους νέους ε, κύκλους δοκιμών που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2017. Πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Ε, και θεωρούμε ότι με όλους αυτούς τους ε, μηχανισμούς θα έχουμε στο μέλλον ε, ένα πολύ καλύτερο οπλοστάσιο που θα ε, μας βοηθήσει και στην πρόληψη αλλά και στην επίτευξη των ε, στόχων για τις εκπομπές που έχουν τεθεί. Κυρία Κρίς Κρόστετ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επανέλθω στην έκθεση του 2013 που μιλούσε για τη διάταξη ε, για την ύπαρξη διατάξεων αλλίωσης. Το είπαν οι συνάδελφοι θεωρούσατε τότε ότι η ύπαρξη τέτοιων συσκευών ε, δεν εντασσόταν στο πεδίο εργασίας της ομάδας, η οποία περιοριζόταν στο θέμα της, των πραγματικών εκπομπών. Διερωτώμε τώρα για την αξιοπιστία των δοκιμών. Μας είπατε ότι χρειάζεται δύο χρόνια πριν να φτάσετε στο πραγματικό δείγμα. Θα έχετε όμως σε συνεχεία εμπιστοσύνη σε αυτές τις δοκιμές. Και τι σύγκριση θα υπάρχει με τις δοκιμές που γίνονται στις ΗΠΑ. Ε, τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα επίσης που προβλέπετε για τα βαρέα οχήματα και τα ελαφρά οχήματα. Um, we've done, uh, quite a lot. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά για να αναπτύξουμε τις ε, διαδικασίες. Ε, μέτρηση εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες, ε, εμπιστευόμαστε το προϊόν μας. Και ε, επίσης υπήρξε μια ερώτηση για τις δοκιμές της ΕΠΑ. Η συσκευή αλλίωσης στις ΕΠΑ στα οχήματα ε, της Volkswagen δεν εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου. Με άλλα λόγια, όλες οι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν στη ΣΥΠΑ δεν εντόπισαν συσκευέ αλλίωσης. Στη δική μας περίπτωση, ε, οι δοκιμές ε, εκπομπών πραγματικής οδήγηση είναι συμπληρωματικές προ τους, προς τις δοκιμές κύκλου. Αν θέλει κανείς λοιπόν να παρακάμψει τους ελέγχους, ε, το κάνει σε αυτή τη φάση και όχι στη, στην, ε, στην άλλη φάση που γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, στο δρόμο δηλαδή. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να παρακολουθεί ολόκληρη την απόδοση της, ε, του κινητήρου. Ε, ώστε να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο, ο κινητήρας είναι καθαρός σε όλες τις συνθήκες. Και για αυτούς τους λόγους είμαστε βέβαιοι ότι το νέο σύστημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε καθαρά οχήματα χωρίς συσκευές αλλίωσης στην αγορά. Και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα θα αποτρέπουμε και την χρήση συσκευών αλλίωσης στο μέλλον. Με βάση αυτά που μας εξηγήσατε για τη σημερινή κατάσταση, ποια είναι η λύση που θα μας επέτρεπε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και το συντονισμό μεταξύ JRC και Κομισιόν, γιατί έχει κάνει την εντύπωση ότι οι πληροφορίες δεν ρέουν όπως πρέπει πάντα. Καταρχήν, εμεί είμαστε Κομισιόν, είμαστε τμήμα τη Κομισιόν, είμαστε υπηρεσία της Κομισιόν. Ασφαλώ το γνωρίζω. Ε, όμως ε, στην Κομισιόν υπάρχουν και διάφορε γενικέ διευθύνσει και οι πληροφορίε θα πρέπει από εσά να φτάνουν να διοχετεύονται στι αρμόδιε ε, γενικές διευθύνσεις. Και έγινε αυτό. Ε, ήταν ενημερωμένοι για τις μελέτες. Ε, για το παρελθόν η πρώτη μου ερώτηση. Μάθαμε σήμερα ότι ε, δεν είναι τμήμα της εντολής σας να είστε φιλίποπτοι. Κάνατε μια προσπάθεια όμως να ενημερώσετε τα κράτη-μέλη για τα πορίσματα των δύο μελετών σας, έτσι ώστε να τα αξιολογήσουν και κάτι για το μέλλον μιλήσατε, είπατε ότι προκειμένου να εντοπίσετε αυτές τις συσκευές παράκαμψης χρειάζεται πρόσβαση στο software. Ε, θα έχετε τέτοιου είδους πρόσβαση στο μέλλον και θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουν τύχη ε, παρέμβαση σε αυτά τα συστήματα στα οποία εσείς θα έχετε πρόσβαση. Ε, τα πρώτο σας ερώτημα για τα κράτη-μέλη πριν την έκθεση του 11 είχαν ε, ενημερωθεί από την Κομισιόν για τα πορίσματά μας μέσω ενός εργαστηρίου που είχε ε, διοργανώσει η Κομισιόν. Και μετά δημιουργήθηκε και η ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν και τα κρατημέλη, ε, εμπειρογνώμονες, μηχανικοί κλπ. Και στις δύο περιπτώσεις οι προσκλήσεις ε, ήταν ε, πολλές, οι συναντήσεις ήταν σχετικά ανοιχτές, ε, δεν περιορίστηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων και επιπλέον στα αποτελέσματά μας εντοπίσαμε διάφορα σενάρια τα οποία αναφέραμε, είχαμε δημοσιεύσει τεχνικά περιοδικά, σε επιστημονικά περιοδικά, συγγνώμη, και πολλά στοιχεία στο site μας. Οπότε επουδενή δεν διατηρήσαμε κρυφές αυτές τις πληροφορίες. Από την αρχή ήμασταν πολύ ανοιχτοί. Δεύτερη ερώτηση, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Ο, κ. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Αν ε, γνωρίζουμε τι κάνει ένα software, ένα πρόγραμμα, είναι σχετικά εύκολο να δοκιμάσουμε το κατά πόσον ε, κάνει αυτό που λέει ότι κάνει. Και με αυτόν τον ε, τρόπο θα διευκολυνθούμε στο να διαπιστώσουμε αν το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται όπως λέει ο κατασκευαστής ότι συμπεριφέρεται. Ε, οπότε δεν μας νοιάζει αν κάποιος έχει παρέμβει στο software ή όχι. Εμείς θα δοκιμάσουμε αν το software κάνει αυτά τα οποία λέει ο κατασκευαστής του ότι κάνει. Οπότε αν έχετε πρόσβαση στο software θα μπορέσετε να εντοπίσετε, θα μπορείτε να εντοπίζετε μια συσκευή παράκαμψης. Ε, ε ελπίζω ότι αυτό θα το, θα το καταφέρουμε και χωρίς πρόσβαση στο software. Ο κ. Ε, Εγώ θα επαναλάβω κάποια πράγματα που είπαν κι άλλοι συναδέλφοι. Είναι ξεκάθαρο ότι το 2013 στην έκθεση υπήρχαν αποδείξει. Ε, έστω και αν λέγονται εδώ ε, ότι υπήρχαν ε, ενδείξει για συσκευέ αλλίωση που μπορούσαν να παραπείσουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή μιλούμε για τη δυνατότητα μια απάτη. Επειδή έβαλαν και άλλοι συναδελφοί και πρόσφατα ο συνάδελφος Ζωρίνιο, δεν απαντήσατε ε, ε, κυρία Κουτέρη, ενημερώσετε την Επιτροπή. Ποιον ενημερώσετε. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ε, η ευθύνη κάθε ερευνητικού κέντρου όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει δυνατότητα απάτης απέναντι στους πολίτες οφείλει να ενημερώσει. Είναι αρμοδιότητα να ενημερώσει ε, πρώτα-πρώτα την Επιτροπή αλλά λέω και τα κράτη-μέλη. Δεν διαπιστώσαμε δηλαδή από αυτά που είπατε ότι ενημερώσατε επαρκώς και σωστά και ποιου ενημερώσατε γιατί το να εξαρτούμαστε σε workshop δεν νομίζω ότι αυτό είναι ενημέρωση ε, και η ευθύνη της, ε, του GRS είναι ε, να ενημερώνει για να μπορεί όπως είπατε πολύ σωστά να πετυχαίνουμε το επίπεδο πρόληψης. Να επιστρέψω σε αυτά που έλεγα. Στην έκθεσή μας εξηγήσαμε για τους λόγους για τους οποίους θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Δεν αναφέραμε ποτέ ότι ένας από τους λόγους μπορεί να είναι αυτές οι συσκευές παράκαμψης. Δεύτερον, Η δουλειά αυτή ξεκίνησε μαζί με την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Κομισιόν. Δεν ξεκινήσαμε με δική μας πρωτοβουλία αυτήν την έρευνα. Πολύ δε περισσότερο που η έκθεση την οποία αναφέρατε, του 2013, ασφαλώς και ήταν εγνώση της Κομισιόν. Ε, ήταν και ένας από τους συντάκτες. Ε, δεν ενημερώθηκαν μέσω του workshop στην Κομισιόν. το, το, το, το σεμινάριο αυτό το είπαμε, το αναφέραμε, γιατί μέσω αυτού ενημερώθηκαν τα κράτη-μέλη. Και σας είπα ότι ήταν μάλιστα και πολύ ανοιχτό. Η Κομισιόν γνωρίζει, γνώριζε την έκθεσή μας, ήταν συντάκτης, ένας από τους συντάκτες, την συγχρηματοδότησε και δεν περίμενε το εργαστήριο αυτό, το σεμινάριο, για να ενημερωθεί. Το σεμινάριο αυτό ε, είχε ευρεία συμμετοχή, ήταν ανοιχτό σε πάρα πολλούς φορείς για να ενημερωθούν αυτοί οι φορείς, όχι οι Κομισιόν. Ενημερώσατε την Κομισιόν, ζητήσατε από τότε, είχετε κάποιες προτάσεις για ανάληψη δράσεων ώστε να διορθωθεί η κατάσταση. Yes, they ναι, όπως σας είπα, η Κομισιόν γνώριζε πολύ καλά τα πορίσματα γιατί ήταν ένας από τους συντάκτες του εγγράφου. Οι δράσεις που αναλήφθησαν ήταν η σύσταση της ε, ε επιτροπης RDLDV στόχος αυτής της ομάδας εργασίας ήταν να βελτιώσουμε τις μεθοδολογίες δοκιμών για να συνεχίσουμε να μειώνουμε τους ρήπους, τις εκπομπές και η ομάδα εργασία αυτή ήταν και πάλι ανοιχτή ευρεία συμμετοχή. Κυρία Ντέλη. Merci. Με μετρήσατε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις εργαστηριακές μετρήσεις και τις πραγματικές μετρήσεις. Αλλά δεν μεταφέρατε αυτές τις προφορίες στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα μοντέλα και τις μάρκες. Ναι, και τις, ε, μάρκες ναι. Ε, ποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Γιατί δεν το κάνατε εσείς. Και από ποιον περιμένατε να το κάνετε. Να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη για συγκεκριμένες μάρκες και μοντέλα. Και δεύτερον, θα μπορούσατε να μου πείτε αν ο Διευθυντής ε, Ενέργειας και Μεταφορών ε, βρίσκεται ακόμα στα καθήκοντά του, επιτελεί τα καθήκοντά του και για ποιο ε, λόγο αναγκάστηκε σε παρέτηση την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπα και προηγουμένως, η, ε, η έρευνα ε, δεν έγινε ε, υποτύπων αστυνόμευσης ε, επειδή θέλαμε να εντοπίσουμε μια συγκεκριμένη μάρκα ε, ή για να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο και γι' αυτό λόγω να ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη. Το πεδίο μας, το πεδίο της έρευνας ήταν η βελτίωση των μεθοδολογιών της, των δοκιμών καταρχήν για τα βαρέα οχήματα και κατόπιν ε, για τα ελαφρά. Το είπα και προηγουμένως ότι ε, δεν έχουμε καθήκοντα στην αστυνόμευσης. Εμείς κάνουμε έρευνα για τη βελτίωση της τεχνολογίας. Για τη μείωση των εκπομπών. Ναι, τα κράτη-μέλη έμαθαν για τα αποτελέσματα. Σας είπα, το σεμινάριο αυτό ήταν ανοιχτό. Τα κράτη-μέλη ήταν εκεί. Η ομάδα εργασίας RDLDV επίσης ήταν ανοιχτή. Κλήθηκαν τα κράτη-μέλη. Και ήρθαν. Το θέμα των μοντέλων και των συγκεκριμένων αυτοκινητοβιομηχανιών. Δεν μα απασχόλησε αυτό στην έρευνά μα. Στην έρευνά μα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε διαφορέ ανάμεσα στο ε, ντίζελ και τη βενζίνη. Και γι' αυτό το λόγο ε, δεν πήγαμε στις ίδιες αυτοκινητοβιομηχανίες για να πάρουμε αυτοκίνητα για την έρευνά μας, αλλά σε εταιρεία νοικίας αυτοκινήτων. Έτσι. Ε, και εδώ είμαι δίπλα σε έναν από τους θυματάρχε μας, τον Αλόης, το ερώτημα το κατά πόσον ο επικεφαλής μια συγκεκριμένη υπηρεσία ε, εξαναγκάστηκε παρέτηση. Δεν εξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Δεν καταλαβαίνω από πού πήρατε αυτέ τι πληροφορίε. Το GRC βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης. και μεσές διευθυντικές τελέχεις και ανώτερες διευθυντικές θέσεις ε, ε, αλλάζουν χέρια ε, το συγκεκριμένο άτομο βρίσκεται στη θέση του. Ε, κοίτα τι τύχη, τι σύμπτωση. Ε, λέει ο κ. Τούρμες. Η κυρία Ντέλη κάνει την ερώτηση. Συγγνώμη κύριε Τούρμες. Δεν έχετε το λόγο. Κυρία Ντέλη, σε συντομία. Θα μπορούσατε να μου πείτε λοιπόν τι ευθύνες έχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο άτομο ποια είναι τα καθήκοντά του. Είναι απίστευτο, λέει ο κ. Τούρμε. Ε, είναι υπεύθυνο για την ενέργεια τη μεταφορέ. Είναι ακόμα υπεύθυνο του Ινστιτούτου του. Κανένας δεν απολύθηκε και στην Κομισιόν υπάρχει το σύστημα της κινητικότητας, ανώτεροι διευθυντικά στελέχη μετακινούνται. Ο κ. Τούρμες λέει κάτι εκτός μικροφώνου. Το GRC ήδη εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική από πέρσι. Ε, κάναμε μια εξωτερική αξιολόγηση του πρόγραμματος της Ρωσία μας και ως τμήμα αυτής της αξιολόγησης μας ζητήθηκε να επανεξετάσουμε την μακρόχρονη στρατηγική μας ένα τμήμα αυτής της στρατηγικής ήταν να ξαναδούμε την εσωτερική μας οργάνωση. Ε, και το κάναμε. Και αυτό το ξεκίνησε πέρσι. Όχι κύριε Τούρμες. Υπάρχει κάποιο θέμα που αφορά την ε, δική μας εργασία. Θα επανέλθουμε. Δεν μου αρέσει το στυλάκι αυτό. Θα σας δώσω το λόγο μια στιγμή. Στη συνάντηση των συντονιστών κάναμε διεξοδικές και σκληρές συζητήσεις, αλλά πολύ σωστές και τελικά συμφωνήσαμε μια μέθοδο εργασίας. Εάν μια πολιτική ομάδα τώρα παρεκκλίνει ε, από αυτό που συμφωνήσαμε, δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν μπορεί ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται έτσι. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα επανέλθουμε στου συντονιστέ. Αν θέλετε να αλλάξουμε την ε, μέθοδο υποβολή των ερωτήσεων κανένα πρόβλημα. Αλλά θα το αποφασίσουμε αυτό στη συνάντηση των συντονιστών. Ναι, ένα διαδικαστικό πρόεδρε. Ζητώ να είσαστε πολύ πιο αυστηροί στην κατανομή του χρόνου. Όλες οι ομάδες έχουν ερωτήσεις και έχουμε και άλλο πάνελ στη συνέχεια. Δεν είναι σωστό μία ομάδα να μονοπολεί το χρόνο και στην πραγματικότητα να μην παίρνει και πληροφορίες. Σας παρακαλώ, δείξτε αυστηρότητα με το χρόνο. Βεβαίω θα το κάνω. Παράλληλα, χρειαζόμαστε μια ε, εξισορρόπηση. Αν προκύψει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, ε, α αφήσουμε λίγο χρόνο για να δοθεί μια απάντηση. Μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την πρώτη ακρόαση. Να δώσω κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Εάν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις, μπορούμε να τις υποβάλουμε γραπτός και θα επαγρυπνήσουμε για να λάβετε απάντηση. Όπως είπα και στην αρχή, θα πάμε στο Ίσπρα, στην Ίσπρα και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να υποβάλουμε ερωτήσεις. Ε, θα πάμε τον Ιούλιο στην Ίσπρα. Τρίτον, όπως είπα και στην αρχή, ζητήσαμε πολλά έγγραφα και ένα από αυτό είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων όλων αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων αυτής της ομάδα εργασίας, κυρίως RDE, LDV, ε, και σε 10-15 μέρες το αργότερο θα έχουμε τα πρακτικά και θα σας τα διαβιβάσουμε. Όπως είδατε, υπάρχουν άπειρες ερωτήσεις, δεν απαντήθηκαν όλες. Θα επανέλθουμε όμως, δεν θα σας αφήσουμε έτσι ήσυχους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και που μας δώσατε κάποιες απαντήσεις. I would like to move to point, um... να πάμε στο σημείο 4, που είναι η επόμενη ακρόαση. Ο κύριος ε, Φράνκο Βιτσέντε θα ήθελα να έρθει στο βήμα, παρακαλώ. colleagues, since Είναι πολύτιμο, συνάδελφοι. Θα ήθελα να περάσουμε στο σημείο 4, την ακρόαση του Διεθνού Συμβουλίου Καθαρών Μεταφορών. Έχουμε όλοι λάβει μέσω email τις απαντήσεις στις ε, γραπτές ερωτήσεις. Υπάρχουν οι απαντήσεις αυτές στο φάκελο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις. Μην τις ξανά Θα ήθελα ο κύριος Φράνκο Βιντσέντε να κάνει μια σύντομη παρέμβαση, 10 λεπτά το πολύ, γιατί, κοιτάξτε, όλα θα επαν... σε όλα θα επανέλθουμε μέσω των ερωτήσεων ούτως ή άλλως. Κυρία Πρόεδρε, ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, λέγομαι Βιτσέντε Φράνκο και είμαι ερευνητής ε, στο Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών. Έχω ειδικότητα στα ελαφρά και βαρέα οχήματα και σε εκπομπέ του. Εκ μέρου του ICCT, με, με τα τιμή συμμετέχω σε αυτή την ακρόαση και με χαρά θα βοηθήσω την Επιτροπή για να συνεχίσει την έρευνά τη ε, για τη μέτρηση και τον έλεγχο των εκπομπών των οχημάτων. Είμαστε ανεξάρτητος οργανισμός, ε, μη κερδοσκοπικός, έχουμε πραγματογνωμοσύνη στα βαρέα και ελαφρά οχήματα, ε, στα καύσιμα, στην αυτιλία, στην αεροπλοεία, στο κλίμα και στη δημόσια υγεία. Θέλουμε να βοηθήσουμε τι ε, υπηρεσίε του δημόσιου τομέα να εφαρμόσουν του κανονισμούς για να μειωθούν οι κλιματικέ αλλαγέ και να βοηθήσουμε την δημόσια υγεία. Ε, το κάνουμε αυτό με, δίδοντας υψηλής ποιότητας στοιχεία που βασίζονται ε, και ανάλυση ε, σημαντική για του πολιτικού και του stakeholders που χρειάζονται έγκαιρα ακριβεί και επίκαιρε πληροφορίε. Οι δημόσιοι φορείς ε, και οι ΜΚΟ με τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε συμπεριλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, προστασίας του περιβάλλοντος, ε, το Συμβούλιο της Καλιφόρνιας για τους αέριους πόρους, ε, το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργεία της Κίνας, την Ιδίας, του Μεξικού και της Βρασιλίας. Επίσης συμμετέχουμε στην παγκόσμια πρωτοβουλία για την εξοικονόμηση καυσίμων, στο συνασπισμό για το κλίμα και το καθαρό αέρα για τη μείωση των βραχίδιων ρηπαντών στις σημερινές μου παρατηρήσεις θα εστιάσω στις πραγματικές εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου, τα νόξ όπως λέμε, που είναι πολύ δύσκολα να ελεγχθούν, ειδικά για τα διζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα. Είναι επιβλαβείς ε, μολυντές αυτοί, ε, αντιδρούν και με άλλες ενώσεις και σχηματίζουν μικρά σωματίδια, καθώς ε, ε, καθώς και όσων στο επίπεδο του εδάφους, ε, που είναι συστατικά του νέφους. Ε, κάνουν κακό στην υγεία, κάνουν κακό στο συστούς των πνευμόνων, μειώνουν την αναπνευστική λειτουργία, προκαλούν αναπνευστικές αρρώστιες, εμφύσιμα και άλλα. Ε, τα αισθάνονται και υγιείς άνθρωποι, αλλά κυρίως οι ευαίσθητοι, όπως είναι όσοι έχουν άσθημα, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόοδο θάνατο οι κινητήρες εσωτερικής καύσης ιστορικά ε, ξέρουμε ότι παράγουν πολλά τέτοια σωματίδια, ε, οξύδια δηλαδή του αζότου, που παράγονται από την αντίδραση αζότου και οξυγόνου κατά τη διάρκεια της καύσης. Οι τεχνολογίες που έχουμε μπορούν να ελέγξουν τις εκπομπές αυτές α, και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες. Αλλά ο έλεγχος αυτών των εκπομπών, ε, ειδικά για διζελοκίνητα, ε, τεχνικά είναι πολύ προβληματικός. Ε, για μελιτέα ωφέλη στην ε, κατανάλωση των καυσίμων, ε, για την βολή των χρηστών και για το κόστος τεχνολογίας, πληρώνουμε ψηλό το τίμημα με τις επιδόσεις των εκπομπών. Τα τελευταία 15 χρόνια τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις εκπομπές των οξυδίων του αζότου για τα διζελοκίνητα αυτοκίνητα έχουν γίνει πολύ αυστηρές. Αλλά ενώ έχουν μειωθεί κατά τη οι πραγματικές εκπομπές, στην πραγματικότητα δεν ακολουθούν ε, την ε, πορεία ε, των όριων που προβλέπει η νομοθεσία. Στην πραγματικότητα, με βάση το σημερινό πρότυπο Euro 6 του 2015, έχουμε ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια που είχαμε πριν από 15 χρόνια στην Ευρώπη με το Euro 3. Εκτιμούμε ότι οι, εκπομπές, οι πραγματικές εκπομπές του, των οξυδίων του άνθρακα αυτά τα διζελοκίνητα αυτοκίνητα ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια 7 φορές είναι το υψηλότατο επίπεδο ε, υπέρβασης από τότε που υιοθετήθηκαν στην Ευρώπη ε, τέτοιες, τέτοιοι κανονισμοί. Η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη γνώριζε τις υψηλές εκπομπές εδώ και πολλά ε, χρόνια, πολύ πριν το 2015. Οι υψηλές εκπομπές συμβαίνουν ε, όταν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή όταν είναι πολύ απαιτητική η οδήγηση, όταν ας πούμε γίνεται ε, ξαφνική επιτάχυνση, όταν ανεβαίνει μια ανηφόρα. Ε, και όμως είναι τμήμα της κανονικής λειτουργίας του αυτοκινήτου και δεν τα, αυτά δεν τα συλλαμβάνει οι, οι εκπομπές, ε, οι δοκιμές έγκρισης τύπου δεν, δεν τα απεικονίζουν καλά, δεν τα πιάνουν αυτά τα στοιχεία. Ε, τότε κάναμε ένα project ε, στην ICCTC σε συνεργασία, το 2013 και 2014 συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής ε, Βιρτζίνια, ε, μαζί με την... Ε, και αυτό, από αυτό το project η, υπηρεσία, η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Αρίων Πόρων της Καλιφόρνιας ανακάλυψαν την χρήση τέτοιων συσκευών παράκαμψης από τη Volkswagen. Κάναμε μια μελέτη του, τον Οκτώβριο του 2014 ε, που έδειξαν ότι έχουμε ξεπεράσει 7 φορές τα όρια του Euro 6. σε πολλές περιπτώσεις ε, η υπέρβαση δεν οφείλονται στην ε, προβληματική οδήγηση, αλλά ε, έχουν να κάνουν με την απότομη αύξηση του φορτίου του κινητήρα, ας πούμε, κάτι που συμβαίνει καθημερινά στην οδήγηση, ή λόγω των συστημάτων επεξεργασίας των καυσαερίων. Αυτή η μελέτη ε, έδωσε αδιάστατα στοιχεία ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συμμόρφωσης ε, με τα πρότυπα για τα οξύδια του άνθρακα. Ε, κάποια από τα οχήματα που ελέγξαμε είχαν όμως μέσα σε εκπομπές κοντά ή κάτω στο, στα όρια Euro 6, αλλά υπάρχουν λοιπόν οι τεχνολογίες, αλλά δεν τις χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές γιατί δεν τους δίνουν αρκετά κίνητρα οι πολιτικές ε, και επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Εδώ σας δίνω και μια γραφική παράσταση της διάστασης του προβλήματος. Επίσης αναλύσαμε και ένα μικρό ποσό α, δεδομένων ε, από φορτηγά ε, επίπεδου Euro 6 και βλέπουμε ότι τα μοντέρνα φορτηγά είναι πιο καθαρά, δηλαδή εκπέμπουν ε, λιγότερα γραμμάρια οξυδίων του αζότου ανά χιλιόμετρο ε, κατά τη διάρκεια τη οδήγηση από ότι τα αντιζελοκίνητα αυτοκίνητα. Κατά την άποψή μα, οι δοκιμέ συμμόρφωση κατά την οδήγηση με τη χρήση των PEMS ε, που χρησιμοποιούνται από, στην Ευρώπη από το 2014 για τα φορτηγά είναι λόγος που συμμορφώνεται τα φορτηγά. Η δικαιομία εν χρήση είναι απαραίτητο στοιχείο οποιασδήποτε αποτελεσματικής ε, στρατηγική για τη συμμόρφωση. Με τον κανονισμό για τι εκπομπέ πραγματική οδήγηση και τι προτινόμενε αλλαγέ στο πλαίσιο τύπου, έγκριση τύπου, η Κομισιόν έχει κάνει ήδη κάποια βήματα για τη βελτίωση των συστημάτων μέτρηση και παρακολούθησης των εκπομπών NOx. Η χρήση δοκιμών εν χρήση για την έγκριση τύπου των επιβατικών οχημάτων είναι μια πρωτοπόρα καινοτομία και οι προτινόμενες διατάξεις για την επιτήρηση αγοράς είναι ε, πολύ σημαντικές. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά. Όπως είπα, η δοκιμή εν χρήση είναι κρίσιμη σημασία στοιχείο ε, μιας αποτελεσματικής ε, στρατηγικής για τη συμμόρφωση. Η επέκταση λοιπόν της επικέντρωσης του κανονισμού RDE πέραν από την έγκριση τύπου στην ε, δοκιμή εν χρήση των οχημάντων που έχουν ληφθεί από ιδιώτες και στόλους θα μπορούσε να ωφελήσει σημαντικά τον έλεγχο των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Η επέκταση των οριακών συνθήκων του, της δοκιμής RDE και η συμπερίληψη των εκπομπών μετά την εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ε, ολοκληρωμένες και ακριβείς μετρήσεις. Η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την δημόσια λογοδοσία και θα πρέπει να δίνονται τέτοιες πληροφορίες στο κοινό που θα αφορούν και την ε, δοκιμή των οχημάτων και μεταξύ αυτών και τους συντελεστές φορτίου κινητήρα. Παρά κάποιες θετικές πλευρές, το προτινόμενο νέο πλαίσιο έγκρισης τύπου δεν υπερβαίνει ή δεν καταφέρνει να αποσαφηνίσει ορισμένες ασάφειες στο ρυθμιστικό πλαίσιο που απαγορεύουν τις ε, συσκευές αλλίωσης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ε, ένα σύστημα, ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής εκθέσεων και εγκρίσεων για τη χρήση ο, ε, οποιασδήποτε εναλλακτική βαθμονόμησης ελέγχου εκπομπών ε, με απέτηση να, να κοινοποιείται η χρήση ή η παρουσία στοιχείου του σχεδιασμού που θα μπορούσε να αλλάξει τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου των εκπομπών του οχήματος κατά την λειτουργία βάσει παραμέτρων όπως είναι η θερμοκρασία, η ταχύτητα, η ταχύτητα του ε, η ταχύτητα που χρησιμοποιείται ε, και ε, θα πρέπει βεβαίω αυτές τις πληροφορίες να έχουν πρόσβαση και ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα. Σας ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο και πάλι πέντε λεπτά η κάθε ερώτηση. Καταρχήν οι δύο συγκητές. Ο κ. Μπιτεκάιν, Θάλπα Μπιτεκάιν. Ε, έχω περιέργεια. Από πού προέκυψε το ενδιαφέρον του, της οργάνωσής σας ε, να εξετάσει το ζήτημα. Κάποιοι λένε ότι επισήμως ή ανεπισήμως η Κομισιόν σας το έθεσε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον σας, έφτασε κάποια πληροφορία μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν όχι, γιατί ξεκινήσατε να ερευνάτε το ζήτημα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο του 2014 ε, αναγνωρίζατε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούσε προηγούμενο για άλλες περιοχές του κόσμου. Για μια και ήταν η πρώτη περιοχή του κόσμου που άρχισε να χρησιμοποιεί τα ε, για την ε, μέτρηση εκπομπών. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ε, συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφενός και των κρατών μελών αφετέρου τη στάση του σε σχέση με αυτό το θέμα. Oh, Να σας απαντήσω με τη σειρά. Ε, το ενδιαφέρον του ICCT για τις πραγματικές μετρήσεις προκύπτει από το γεγονός ότι είμαστε μέλη της ερευνητικής κοινότητας. Είμαστε ερευνητέ. Και ήταν γνωστό ότι αυτό ήταν ένα εκρεμές ε, θέμα. Ένα ανοιχτό θέμα. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ε, ήταν ε, επίκαιρο ε, ερευνητικό ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να εργαστούμε. Γι' αυτό δεν ε, το έθεσε υπόψη μας η Κομισιόν. Δεν χρειαζόταν κιόλα, μια και υπήρχαν αρκετά ε, ερευνητικά papers, ερευνητικέ εργασίε οι οποίες είχαν δημοσιευθεί και είχαν ελεγχθεί από άλλου ερευνητέ, οπότε ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε, δεν χρειαζόταν να μας ενημερώσει. Ε, άλλωστε η Κομισιόν δεν αποφασίζει για το τι θα ερευνήσουμε και τι όχι, ήμασταν εξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα. Μετά αναφερθήκατε στην έκθεση του Οκτωβρίου 2014, όπου αναφέρουμε ότι η Κομισιόν έκανε πολύ καλή δουλειά. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, grand trabajo είπατε στα ισπανικά, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι αυτό αναλέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, πράγματι επενέσαμε την ε, Κομισιόν που ξεκίνησε την ε, ομάδα εργασία το 2011 και πράγματι ήταν πρωτοπόρα η χρήση των PEMS στην μέτρηση των πραγματικών εκπομπών. Οπότε καλά κάναμε και επενέσαμε την Κομισιόν. Ο έπαινος της άξιζε. και σε ό,τι αφορά την, γνώση, την άποψή μου για την στάση της Κομισιόν και των κρατών μελών. Από πότε? Από το 2011 ή από το 2015? Και τα δύο. Οπότε να ξεκινήσω από το Σεπτέμβριο 2011. Πιστεύουμε πως η Κομισιόν προέβηκε σε σωστή διάγνωση, ακόμα και πριν εμφανιστεί ασθένεια, πριν το πρώτο κρούσμα. Αν δείτε το, χρονισμό της, ε, των, της εμπορίας των οχημάτων γύρω 6, ξεκίνησε το 2011 και μάλιστα με πολύ μικρή με πολύ μικρά νούμερα. Νομίζω ότι σχεδόν καθόλου ε, δεν πωλήθηκαν το 2011, κάποια λίγα μοντέλα το 2012. Η Κομισιόν από το 2011 εντόπισε ότι θα υπήρχε θέμα εφαρμογής του νόμου, εκτός και αν ελαμβάνονται μέτρα. Και γι' αυτό το λόγο άρχισε να μιλά για ε, μετρήσεις, πραγματικές μετρήσεις ε, κατά τη διάρκεια της χρήσης με τυχαίους ε, κύκλους ελέγχου. Τότε βέβαια δεν είχε στο μυαλό της τόσο πολύ η Κομισιόν το θέμα των διατάξεων παρά, παράκαμψης, αλλά ε, πιο πολύ το θέμα του κύκλου ο οποίος ε, χρησιμοποιείται στα εργαστηριακά ε, στις εργαστηριακές ε, δοκιμές ε, ο οποίος προβλέπει μικρό φορτίο ενώ αντίθετα οι εκπομπές οξυδίων του αζότου αυξάνονται εκθετικά όταν το φορτίο αυξάνεται οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε και υψηλές εκπομπές ακόμα και απουσία τέτοιων διατάξεων παράκαμψη. Επόμενη ερώτηση ο κ. Γεμπράντη τρεις ερωτήσεις όπως είπατε πολύ ξεκάθαρα στην παρουσίασή σας, η υπέρβαση ε, των ορίων διοξιδίου των, οξυδίων των αζωτών δεν είναι κάτι καινούριο. Ο ICCT το μελέτησε αυτό και πριν το 2013 ή μόνο από το 2013 και μετά το αρχίσατε να το εξετάζετε. Δεύτερον, διαφορά ανάμεσα στα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Νομίζω ότι μία από τις βασικές διαφορές είναι ότι στην Ευρώπη οι δοκιμές ε, δημοσιεύονται. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι μυστικό το πώς δοκιμάζουν τα οχήματα. Ποια από τις δύο μεθόδους πιστεύετε ότι είναι πιο δίκαιη ε, και καθιστά πιο εύκολη την παρακολούθηση και την εφαρμογή του νόμου. Τρίτον, στις γραπτές σας απαντήσεις, στην απάντηση της ερώτηση 3, λέτε ότι οι διατάξεις παράκαμψης μπορούν να εντοπίσουν πιστούν με τις υπάρχουσες ε, μεθόδους και τα, τα υπάρχοντα όργανα. Το JRC από την άλλη μεριά λέει ότι δεν είναι δυνατόν με την σημερινή τεχνολογία κάτι τέτοιο. Χρειάζονται πολύ πιο προχωρημένες μεθόδους, αναλυτικές μεθόδους και δεν έχουν την δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Εσείς όταν λέτε ότι οι μέθοδοι που έχουμε και τα μέσα που διαθέτουμε είναι επαρκή ε, για τον εντοπισμό. Αυτός ο εντοπισμός θα ήταν πολύ ακριβώς, ε, θα μπορούσε να γίνει με οικονομικό τρόπο. Ευχαριστώ. Thank you. Ναι, ε, η, τα οξύδια του αζότου είναι κάτι καινούριο και η υπέρβαση το ICCT νομίζω ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για βαρέα οχήματα πιο πολύ για αυτό το ζήτημα και μπορώ να σας πω ότι και εγώ προσελήφθη το 2013 ειδικά για αυτό το θέμα. Το 50% του χρόνου μου έπρεπε να αφιερωθεί ερευνητικά σε αυτό το ζήτημα. Αυτό προέβλεπε η σύμβασή μου. Τελικά αφιέρωσα το 90%. Γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον, είχαμε πολλά να κάνουμε. Μιλώ για το 2013 βέβαια. Οπότε ναι, είχε γίνει κάποια δουλειά, αλλά για τα βαρέα οχήματα πιο πολύ από τον ICCT πιο πριν. Ε, λέτε ότι στις ΗΠΑ ε, ε, δεν γνωρίζουμε πώς γίνονται οι δοκιμές. Οι στις ΗΠΑ εφαρμόζεται η δοκιμή chassis, dyno, με πολλαπλούς κύκλους. Εσείς ε, μιλάτε πιο πολύ για μια καινούργια προσέγγιση των ε, αρχών των ΗΠΑ, του EPA κλπ, ε, η οποία ξεκίνησε μετά το σκάνδαλο. Έστειλαν μια επιστολή στις αυτοκινητοβιομήνες και τις ενημέρωσαν ότι από εδώ και πέρα οι δοκιμές θα γίνονται με PEMS, τυχαίους κύκλους, αισθητήρε εξ αποστάσεω κλπ, Ένα σύστημα το οποίο δεν περιγράφεται πολύ. Καλό αυτό. Αυτό δεν αφορά την πιστοποίηση, την έγκριση τύπου, όσο την, τον εντοπισμό των ε, διατάξεων παράκαμψης. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό γιατί εισάγει ένα στοιχείο τυχαιότητας. Δεν θέλουν να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοναδικό πρωτόκολλο στην ε, στον εντοπισμό των διατάξεων παράκα, ε, παράκαμψης ε, χρειάζεται κανείς να έχει μια σειρά, ένα οπλοστάσιο εργαλείων και όχι μόνο ένα πρωτόκολλο, γιατί ένα πρωτόκολλο δεν λειτουργεί από μόνο του. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει σωστά, λειτουργεί σωστά. Χρειάζεται να έχουμε ένα στοιχείο τυχαιότητας, γιατί κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι ψάχνει, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα λειτουργεί η διάταξη την οποία θα εντοπίσει. Έχω χρόνο? Ωραία. Ε, είπαμε ότι οι διατάξεις αυτές μπορούν να εντοπιστούν με τις, χίουσες, με, ε, τις υπάρχουσες μεθόδους και μέσα. Ε, πώς να το ερμηνεύσουμε αυτό. Να σας πω. Ε, θέλαμε να νομίζαμε ότι ρωτούσατε αν περιμένουμε κάποια καινούργια εφεύρεση που θα μας βοηθήσει ή αν χρειάζεται κάποια καινούργια εφεύρεση. Και εκεί απαντήσαμε πως όχι, δεν χρειάζεται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε PEMS, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αισθητήρε εξ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχαίους κύκλους. Τα εργαλεία που έχουμε και οι μέθοδοι που διαθέτουμε είναι επαρκείς για να γίνει ο εντοπισμός. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι εύκολο ή πως γνωρίζουμε πολύ καλά πώς πρέπει να γίνει αυτό. Ε, είναι, είναι δύσκολη επειδή είναι δύσκολο ο εντοπισμό αυτών των διατάξεων, αλλά δεν χρειαζόμαστε παραπάνω εργαλεία. Δεν χρειάζεται κάποια καινούρια τεχνική την οποία δεν διαθέτουμε ε, εύκολα αυτή τη στιγμή. Κύριος Κάνης. Ευχαριστώ. Διάβασα την έκθεσή σας, τη μελέτη σας που το Θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό που είπατε στη σελίδα 5 που αφορά την σύνοψη των όσων αναφέρονται στην σελίδα 3 της μελέτης σας και βεβαίως καθένας μας ε, ενδιαφέρεται ε, προφανώς για ε, τη μη συμμόρφωση. Θέλω να σας ρωτήσω για το όχημα που συμμορφούνται. Υπάρχει όχημα το οποίο σε πραγματικές συνθήκες ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Και το ερώτημά μου είναι εντυπωσιακό. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι μικρός ο κινητήρας, είναι μεγάλος ο κινητήρας. Τι τελικά χαρακτηριστικά έχει αυτός ο κινητήρας αυτού του κατασκευαστή, που του δίνει τη δυνατότητα να συμμορφώνεται. Είναι προφανές ότι η τεχνολογία... Είναι προφανές ότι η τεχνολογία υπάρχει τι κάνουν τελικά αυτοί οι κατασκευαστές που καταφέρουν και συμμορφώνονται. Τι μπορείτε να μας πείτε. Yeah, so that's one car out of 15, uh, unfortunately, like you said. Μπορώ να σας πω ποιος κατασκευάζει το συγκεκριμένο όχημα αργότερα. Αλλά πάντως αυτό που είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο για τα PEMS είναι ότι κάθε φορά έχεις κάτι, κάτι διαφορετικό. Μπορεί να ε, ε, κάνεις διαφορετική οδήγηση και έτσι να λάβεις διάφορα στοιχεία ε, από τις εκπομπές. Σε εμάς τους ερευνητές ε, αρέσει αυτό. Εμείς δυστυχώς έχουμε μόνο δεδομένα μίας ώρας από έναν ερευνητή, από ένα εργαστήριο που έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο κατασκευαστής αυτός δεν αναφέρεται στην ίδια την έκθεση αλλά επειδή ε, ο ίδιος οργανισμός περιβαλλοντικής προστασίας ε, ανέφερε την BMW ε, και την ε, Volkswagen είναι κάτι που μπορεί κανείς να το, να το παρακολουθήσει αν θέλει. Άρα είναι η BMW. Πρόκειται για ένα ε, μοντέλο μεγάλο σχετικά. Στην Ευρώπη έχουμε κίνητρα προς τους αγοραστές να αγοράζουν μικρού κυβισμού αυτοκίνητα με μικρούς κινητήρες. Αυτό είναι τελικά αυτό το μοντέλο είναι μεγάλο ε, και μήπως τελικά αυτές οι, αυτά τα κίνητρα που δόθηκαν στην Ευρώπη για την αγορά μικρών οχημάτων είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Είναι το BMW 3 G3, GT, G3 G20. Είναι μεγάλο αυτό το όχημα. Νομίζω ότι είναι σειρά 3 ε, με μεγάλο προπαγκάζι. Εμένα μεγάλο μου φαίνεται. Ναι, εντάξει, μεγάλο σε μέγεθο. Ο κινητήρα είναι πιο ισχυρό. Νομίζω ότι είναι δίλητρο ο κινητήρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρο, θα επανέλθω. Ε, είναι αλήθεια πάντως ότι, ότι υπάρχει τάση για μικρότερους κινη, τήρες στην αγορά και στην έκθεσή μας του Σεπτεμβρίου 2015 ε, ε, Φαίνεται ότι υπάρχει μία ε, τάση υπέρ των κινητήρων LNT. Άρα λέτε ότι τα κίνητρα που δόθηκαν στους καταναλωτές να αγοράζουν ε, μικρότερους κινητήρες τελικά ήταν ένα μέτρο αντιπαραγωγικό και αύξησαν τις εκπομπές οξυδίου του αζότου. Άρα λέτε ότι οι πολιτικές που χαράξαμε είχαν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Όχι. Λέω ότι η τεχνολογία στα μικρότερα αυτοκίνητα κάποιες φορές είναι χειρότερες. Δηλαδή τα μικρά αυτοκίνητα έχουν μεγαλό μεγαλύτερες, υψηλότερες εκπομπές οξυδίων του αζότου. Ε, κοιτάξτε, ε, είναι, μια πολύ, είναι μια γενίκευση αυτή και δεν μπορώ να, να κάνω μια τέτοια δήλωση. Πάντως με, με τουρμποκινητήρες ε, θα πρέπει κανείς να συνεκτιμά και το, το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι μια γενικότερη ε, διαδικασία και για ένα θέμα που αφορά την γενικότερη κατασκευή των κινητήρων. Ευχαριστώ Κύριε Φράνκο. Καλή απάντηση που, που μου δώσατε ε, στην απάντηση 6 για το διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012. Τώρα, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Καταρχάς, στην ε, ερώτησή σας τρία για τους διάφορους χειρισμούς και τις απάτες. Μου λέτε κάτι ενδιαφέρον. Υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία για να ανακαλύψουμε τις λαθροχειρίες. Αλλά είναι δύσκολο με τους κανόνες που έχουμε σήμερα να διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτό που είναι νόμιμο και σε αυτό που είναι παράνομο. Κατάλαβα καλά. Το πρώτο τμήμα της απάντησης αφορά τα όργανα. Δηλαδή μπορείς να ανοιχνεύσεις μια συσκευή αλλίωσης. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι ψάχνεις καταρχάς και αν ας πούμε η βαθμονόμηση κάποιων συστημάτων καθαρισμού των καυσαερίων είναι τέτοια συσκευή αλλίωση ή όχι. Αν υπάρχει έλλειψη αφήνεια ή αν υπάρχει αμφισημία στον κανονισμό, δηλαδή θέλουμε ένα κανονισμό πιο σαφή, αυτό θέλετε να μα πείτε, διακόπτει ο μιλητή. Χρειάζονται περισσότερε περισσότερες Υπόθηκε πολύ σωστά ότι χρειαζόμαστε κριτήρια αξιολόγηση από κάποιον. Πολύ σωστό αυτό. Και είπατε ότι και η Κομισιόν εργάζεται από αυτό. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν περιγραφές των συνθήκων, των υπό, τον, υπό τις οποίες η εναλλακτική βαθμονόμηση, ας μην τα πούμε συσκευές αλλίωσης, είναι επιτρεπτό και τεχνικά στοιχειοθετείται. Υπάρχουν τα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχουμε τέτοια έγγραφα στην Ευρώπη. Δηλαδή, τα σχέδια, ε, τα σχέδια αυτά των ε, αυτοκίνητων να χρειάζομαστε. Ποια σχέδια του κινητήρα, λέει ο μιλητής. Γιατί αυτό το αναφέρεται και στο σημείο 5.2. Τον, ε, αναφέρεται μάλλον στους ευρωπαϊκούς κανόνες, το σημείο 5.2. Δηλαδή, για να δούμε πώς λειτουργεί ο κινητήρας, χρειαζόμαστε τα σχέδια του κινητήρα. Α, σε αυτό αναφερόσασταν. Ε, μιλάτε δηλαδή για τις εξαιρέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται να έχουμε τέτοιες συσκευέ αλλίωσης στο βαθμό που χρειάζονται για να προστατεύεται ο κινητήρας. Θα πρέπει τεχνικά να δικαιολογείται αυτό. Γιατί αλλιώς, εάν δεν υπάρχει σαφής ορισμός του πότε αυτές οι εξαιρέσεις χορηγούνται, τότε μπορεί να εφαρμόζονται συνέχεια οι συσκευέ αυτές και, αφή, και ανοίγεται το, την πόρτα ορθάνυχτη για λαθροχειρίε, για απάτες κτλ. Θα πρέπει αυτό το παραθέακι να το κλείσουμε, αυτήν την κακόπορτα. Πολύ σύντομα. Είσαστε πάρα πολύ αυστηροί για τους διζελοκινητήρες. Η, μετάβαση προς υβριδικούς κινητήρες είναι εφικτή με, την, με τους διζελοκινητήρες. Εμείς δεν έχουμε καμία προτίμηση προς την τεχνολογία. Μας ενδιαφέρει καθαρή τεχνολογία. Δεν έχουμε πρόβλημα ε, με το ντίζελ αυτό καθεαυτό. Θέλουμε να είναι καθαρό το ντίζελ. Αν είναι βρώμικο έχουμε πρόβλημα όμω. Και μπορεί στο, στο μέλλον ας πούμε, να είναι τμήμα του μείγματο της τεχνολογίας. Δηλαδή το ντίζελ να παραμείνει. Εγώ θέλω να καταλάβω καλύτερα. Φυσικά υπάρχουν ε, βρώμικα και καθαρά ντίζελ, δίζελοκινητήρε δηλαδή. Μια και είμαστε σε φάση μετάβαση, σε μεταβατική φάση προ υβριδικού κινητήρε. Σε αυτή τη ε, μεταβατική φάση είναι καλύτερο να έχουμε δισελοκινητήρε ή βενζινοκινητήρε. Μπορεί να έχετε και τα δύο. Αλλά δεν έχει νόημα να έχετε υβριδικά διζελοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι πιο ακριβό. Το επιπλέον κόστος για την επεξεργασία των καυσαερίων καθιστά το αυτοκίνητο πολύ ακριβό. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια υβριδικά διζελοκίνητα αυτοκίνητα και ο λόγος είναι οικονομικός. Έτσι, είναι πολύ ακριβά. Τελευταία ερώτηση. Εσείς δουλέψατε και στο Ίσπρα και μετά πετάξατε στην Αμερική. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Τελικά είχατε μεγαλύτερη τύχη, ας πούμε, στην Αμερική. Είχατε περισσότερη ελευθερία, περισσότερες δυνατότητες. Όχι, δεν δουλεύω στην Αμερική εγώ, δουλεύω στο Βερολίνο. Είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Δεν δουλεύεις για την κυβέρνηση. Είναι τελείως διαφορετικό να δουλεύεις για ένα ΜΚΟ, ας πούμε, ως ερευνητής. Υπάρχουν κοινά στοιχεία στη δουλειά, αλλά δεν καταλαβαίνω και πού το πάτε. Έχω δουλέψει πάντως και για τις δύο, τους δύο οργανισμούς, ας πούμε. Μία ερώτηση για τις συσκευέ αλλίωση. Ε, και το πώς χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Η δουλειά που κάνει το ICCT ήταν σημαντικό, ούτως ώστε να καταλάβουν οι Αμερικανικέ αρχές ότι χρησιμοποιούνται τέτοιες συσκευέ ε, μέσω των εργασιών που έκανε στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια. Ε, και το εντοπίσαμε το, αυτή τη συσκευή λόγω του ότι είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα με τα PEMS και στο εργαστήριο. τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη. Το SCT έχει εμπλακεί και ακούσαμε ότι υπάρχει ένα μακρύ ιστορικό διαφορών ανάμεσα στις πραγματικές ε, εκπομπές που μετράμε με τις φορτές συσκευές και στις ε, εκπομπές που μετράμε κατά την, ε, τις δοκιμές έκρησης τύπου. Μπορούμε να συνάγουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιήθηκαν ή ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν στην Ευρώπη τέτοιες συσκευέ αλλίωσης. Όταν μιλάμε για συσκευέ αλλίωσης στην Ευρώπη, φαντάζομαι ότι εννοείται υπό ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά ο νόμος στην Ευρώπη και στις ε, είπα. Στην ε, Ευρώπη έχουμε υψηλέ ε, εκπομπέ οξυδίων του αζότου. Τώρα, αν αυτό οφείλεται σε συσκευέ αλύσωση, δεν μπορώ να το πω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η έρευνά σα στι ΗΠΑ ε, κατέδειξε αυτόν τον συσχετισμό και στη συνέχεια η Αμερικανική κυβέρνηση αποκάλυψε την, την όλη ιστορία. Άρα, μήπως η, έρευνά σα καταλήγει σε κάτι παρόμοιο ε, και στην Ευρώπη και τι έχουν κάνει οι διοκτικές αρχές ή οι αρχές ελέγχου, οι ελεγκτικές αρχές στην Ευρώπη. Όταν λέτε, ε, ε, αναφέρεστε στο, στην έρευνα του Πανεπιστημίου της, της Δυτικής Βιρτζίνιας να το διευκρινίσω. Εμείς δεν ε, βρήκαμε συσκευή αλλίωσης. Εμείς αυτό που βρήκαμε ήταν μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των εκπομπών οξυδίων του αζότου και των πιστοποιημένων επιπέδων. Και ήταν πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Γιατί οι εκπομπές εν χρήση ε, ε, ειδικά στην Αμερική ε, είναι πάρα πολύ υψηλές οι εκπομπές στα οχήματα και οι, οι εκπομπές αυτές μετρήθηκαν σε κύκλο που ήταν πιο απαιτητικός από αυτό που προβλέπεται στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνω αυτό λέει, αλλά παρόλα αυτά υπήρξε ένας συσχετισμός ότι ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η διαφορά άξιζε τον κόπο να ελέγξει κανείς μήπως χρησιμοποιήθηκαν συσκευές αλλίωσης. Και εντάξει, ε, ανεξάρτητα από το αν ήταν το ICCT ή το Πανεπιστήμιο της Δυτικής ε, Βιρτζίνιας. Εγώ αυτό που ρωτάω είναι αν κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να είχε γίνει και στην Ευρώπη. Και αν θα μπορούσαμε δηλαδή να συμπεράνουμε ότι αυτού του είδους οι διαφορές οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα στη χρήση συσκευών αλλίωσης. Είναι ειλικρινή η ερώτηση αυτή. Ε, πριν από το σκάνδαλο Volkswagen δεν είχαμε μεγάλα ε, ερευνητικά προγράμματα για τις συσκευέ αλλίωση. Είναι καινούριο πράγμα. Είναι ένα καυτό θέμα πράγματι αυτή τη στιγμή, αλλά ε, το οποίο ανέκυψε μόλις το Σεπτέμβριο του 2015. Άρα στην έρευνά σας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας βοηθήσει να ε, διαπιστώσουμε αν χρησιμοποιήθηκαν συσκευές αλλήλωσης στην Ευρώπη ή όχι. Φαίνεται ότι υπάρχουν ε, πολύ υψηλέ εκπομπές οξυδίων του αζότου σε κάποια οχήματα. Αλλά για να ε, ε καταλήξει κανείς στο ότι χρησιμοποιήθηκαν συσκευές αλλήλωσης χρειάζονται μεγάλες έρευνες. Αυτές οι έρευνες στις ΕΠΑΞ έχουν ξεκινήσει και διαρκούν ακόμη από το 2014. Οπότε είναι πολύ δύσκολο δύσκολο μια ΜΚΟ να κάνει ε, αυτό το έργο. Οι αρχές θα πρέπει να το κάνουν. Εγώ δυστυχώς μηχανικός δεν είμαι, αλλά καταλαβαίνω ότι από αυτές τις υποψίες που προέκυψαν από τα δεδομένα, θα ήθελα να μάθω αν το ICCT έχει να κάνει προτάσεις για το τι θα πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν τελικά χρησιμοποιήθηκαν συσκευές αλλίωσης. Ε, κάτι που δεν σχετίζεται ακριβώς με αυτό που ρωτάτε, αλλά θα δημοσιεύσουμε το δεύτερο κομμάτι της μεταανάλυσης μας και εκεί θα καλύπτουμε 30 τόσα αυτοκίνητα ε, και θα δώσουμε πολύ λεπτομερή στοιχεία. Και θα δημοσιεύσουμε πίνακες που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από πού έχουν προέλθει οι υψηλέ εκπομπές. Θα είναι πάρα πολύ λεπτομερής αυτή η, η έκθεση. Πότε, ε, ρωτάει η Πρόεδρος, ε, θα χρειαστούμε λίγους μήνες ακόμα. Ευχαριστώ. Ε, οι μελέτες σας δείχνουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε ε, μετρήσεις εργαστηριακές και πραγματικές, μετρήσεις πραγματικές συνθήκες στα οξύδια του αζότου. Εφτά φορές περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες. Ε, Για αυτό το λόγο χρειάζονται δεχομένω ε, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Είναι ταυτόχρονα και επιβεβαίωση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο παράγοντας ε, συμμόρφωση θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ ψηλότερα από το 2. Thank uh, ένα σχόλιο για τους μέσους όρους. Είναι πράγματι ο μέσος όρος 7, 7 ε, οι πραγματικές ε, εκπομπές, ε, αλλά υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα, υπάρχουν μοντέλα που έχουν πολύ μεγαλύτερες διαφορές, πολλαπλάσιες του 7. Με την σημερινή τεχνολογία είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με το γύρο 6 σε συνθήκες δρόμου. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμος ένας υψηλός ε, συντελεστής ε, ε, συμμόρφωσης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την τεχνολογία μας. Ε, και εμείς ε, βλέπουμε τα αποτελέσματά μας ως επιβεβαίωση της ανάγκης χρήσης ε, μετρήσεων σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό που συμπεράναμε και εμείς ήταν πράγματι ότι η Κομισιόν είχε δίκιο το 2011 όταν ξεκίνησε την διαδικασία με τα PREMS και ότι χρειάζεται ε, να προβούμε σε μετρήσεις πραγματικών εκπομπών και μάλιστα ακόμα πιο προχωρημένων από αυτές που έχουμε. Ωραία. Κυρία Κιλιόμ. Η κυρία Κιλόναν, συγγνώμη. Έχω μια σειρά ερωτήσεων. Για ποιο λόγο υπό τις παρούσες συνθήκες ε, μάλλον ποιο θα ήταν το κόστος εντοπισμού συσκευών παράκαμψης υπό τις σημερινές συνθήκες. Θα μπορούσαμε να ε, έχουμε επαναλαμβανόμενα πειράματα, επαναλήψιμα πειράματα με PEMS και για τα σωματίδια. Τρίτον, το σύστημα παρακολούθησης του ίδιου του αυτοκινήτου θα μπορούσε να μετρά τις εκπομπές καλύτερα ε, από τη σήμερα. Τε, τελευταίο, τέταρτον, πώς ε, με μετρήσεις ε, εκ των υστέρων μετά την πώληση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουμε ε, την ύπαρξη ε, διατάξεων παράκαμψης. Επαναλαμβάνονται αυτή η ερώτηση. Μετρήσεις μετά την πώληση θα μπορούσαν να εντοπίσουν περισσότερες και άλλες εταιρείες που είχαν χρησιμοποιήσει διατάξεις παράκαμψης. Εννοείται μέσω έρευνα στην αγορά, έτσι δεν είναι. Αυτό εννοείται. Μάλιστα, απάντηση. Για ποιο λόγο να έχουμε ε, διατάξει παράκαμψης. Ο λόγος, όπως το είπα και στην αρχή, είναι ότι ε, για παράδειγμα η τεχνολογία LNT χρειάζεται αναγέννηση του καταλήτη, κάτι που αυξάνει κατά 2-4% την κατανάλωση ε, καυσίμου. Ε, επίσης, αν χρησιμοποιούμε ουρία γενναιόδωρα τότε ε, μειώνεται μειώνονται, μειώνεται η περίοδος ε, γεμίσματος ε, της ουρίας, το οποίο σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να πηγαίνει στο συνεργείο πιο συχνά. Οπότε είναι θέμα ε, ε βολής του ίδιου του καταναλωτή, ευκολίας του καταναλωτή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, το κόστος εντοπισμού αν αυτοκίνητο ε, μπορεί να είναι πολύ χαμηλός αν θέλουμε μια πρώτη ένδειξη και αν έχουμε μια τέτοια ένδειξη, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση, να ακολουθήσουμε μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση για τον πραγματικό εντοπισμό, δεδομένη λέω μια πρώτη υποψία, που θα είναι όμω πολύ ακριβότερη. Εξαρτάται πόσε δοκιμέ θέλουμε να κάνουμε. Ε, τώρα, εντο, ε, μέτρηση σωματιδίων. Τα όργανα μας δεν είναι ε, αρκετά όρημα γι' αυτό. Αλλά α, άκουσα τελευταία ότι μέχρι το 2019 θα μπορούμε να μετράμε και τα σωματίδια. Καλό νέο αυτό. Τώρα, αν τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να μετρούν τις, δικα... τις εκπομπές τους, μόνα τους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ε, αισθητήρε ε, οξυδίων του αζότου και μετρούν τις εκπομπές τους. Νομίζω ότι τα αυτοκίνητα ήδη μπορούν να μετρούν με αρκετή ακρίβεια τις εκπομπές τους. Το θέμα είναι εμείς μπορούμε να εμπιστευτούμε τις μετρήσεις ενός αυτοκινήτου. Παρακαλώ πολύ μην μου θέσετε αυτό το ερώτημα, δεν μπορώ να το απαντήσω. Ε, ίσως ναι, αν μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσουμε επισήμως ε, τα συστήματα αυτά που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα και να τα πιστοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Τελευταία ερώτηση. Είναι πιθανό καινούριες ε, ε διατάξεις ε, παράκαμψης να εντοπιστούν. Δεν, γνωρίζω, όχι θα έλεγα, δεν είναι πιθανό. Δεν, μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει αύριο όμως. Κυρία Άρμς. I would like to ask Να θέσω ένα ερώτημα. Για την πρώτη απάντηση που δώσατε, την πρώτη γραπτή απάντηση στις ερώτηση που είχαμε προϋποβάλει. Μας λέτε σε αυτήν την πρώτη απάντηση ότι παρουσιάσατε τα πορίσματά σας στην πρώτη έκθεση και εκεί μιλούσατε για τις ε, διαφορές ανάμεσα στα όρια που προκλέπει νομοθεσία και στα, σε αυτά που προκύπτουν τις μετρήσεις. Μας είπατε ότι σε μια ομάδα εδώ εργασία στις Βρυξέλλες, παρουσιάσατε τα πορίσματά σας στις 31 Μαρτίου του 2014 και αργότερα τον Οκτώβριο δημοσιεύσατε τη μελέτη σα. για αυτέ τι διαφορές. Και μάλιστα τα αναρτήσατε αυτά στοιχεία και στην ιστοσελίδα σας. Μετά από αυτές τις συζητήσεις και τις δημοσιεύσεις που έλαβαν χώρα και στην ιστοσελίδα σας λοιπά. Οι εθνικές αρχές σας πλησίασαν ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας πλησίασε για να μάθει περισσότερα. Ίσως λίγο πριν ή λίγο μετά, αλλά τη στιγμή που παρουσίασα τα προκαταρτικά μου πορίσματα στην ομάδα RDE LDV το Μάρτιο του 2014 ε, συζητήσαμε τον Κλάου Στάνιγκερ που είναι ο υπάλληλο υπεύθυνο για το RDE και ήρθαμε σε επαφή εδώ, ήρθε σε επαφή με το δικό μα γραφείο στο Βερολίνο. Δεν έχω πρακτικά τη ε, συζήτηση. Αλλά το συμπέρασμα ήταν ότι χρειαζόταν το RDE, δηλαδή οι πραγματικές εκπομπές, και τα αυτοκίνητα που είχαν πιστοποιηθεί στο εργαστήριο μόνο, τελικά δεν ε, είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν μια δοκιμή RD. Αυτά μετά από συζητήσεις με, την, ε, με Γενικής Διεύθυνσης ε, GROW. Θέλω να ψάξω να βρω τον Λίποντα λοιπόν, Κρίκο τεχνολογίας και επιστήμης, αρχών και πολιτικής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία του Περιβάλλοντος, η ΕΠΑ, η Αμερικανική, συγγνώμη, ναι, ε, έδρασε πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί οι ΜΚΟ είχαν δώσει στις αμερικανικές αρχές καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία για τα προβλήματα που υπήρχαν. Το θέμα είναι αν τα αποδεικτικά στοιχεία που δόθηκαν στις ευρωπαϊκές αρχές, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στις εθνικές αρχές, ήταν πιο φτωχά σε σχέση με αυτά που εσείς δώσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Αμερικανικές Αρχές, στην ΕΠΑ δηλαδή, στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η έκθεση που δημοσιεύσαμε το Μάιο του 2014 που πήρε το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια και της EPA και που πήρε και η EPA ε, ήταν μια έκθεση που είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και δεν ναι, την έχουμε κατεβάσει. Η ευρωπαϊκή μελέτη ε, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2014 ήταν λιγάκι διαφορετική γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν ζητήσαμε άμεσες μετρήσεις αλλά συλλέξαμε δέσμες δεδομένων από stakeholders της ομάδας RD και δημοσιεύσαμε ε, σορευτικά αποτελέσματα σε αυτή τη μεταμελέτη. Η διαδικασία είναι λιγάκι διαφορετική αλλά το περιεχό... και το περιεχόμενο ήταν διαφορετικό. Όταν μιλάτε για τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και στην έρευνα, ε, με χαρά και τιμή είμαστε τμήμα αυτού του κύκλου και το JRC είναι. Δηλαδή, λέτε τελικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία με βάση τις προφορίες που προσκομίσατε εσείς, όπως και η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασία του Περιβάλλοντος. Ίδια στοιχεία είχαν και η Επιτροπή και η ΕΠΑ. Για ποια στοιχεία μιλάτε? Το, γραφείο, το κέντρο στο το ICCT, έδωσε τα ίδια στοιχεία στις ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές και στις αμερικάνικες αρμόδιες αρχές. Ε, στην περίπτωση των, της EPA, της Αμερικάνικης εταιρείας, ε, τα στοιχεία που είχαν αφορούσαν ε, πιστοποιημένα αυτοκίνητα στην Αμερικανική αγορά. Είναι τελείως διαφορετικό το context. Η κυρία Εύη. Να επανέλθω στις συσκευές αλλίωσης εγώ. Από αυτά που υπόθηκαν από το ερευνητικό κέντρο, ο εντοπισμός αυτών των συσκευών είναι σχεδόν αδύνατος, εάν δεν μας το πούν οι κατασκευαστές. Περίεργο μου φαίνεται εμένα, βέβαια. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν τεχνικές προϋποθέσεις ή τεχνικοί λόγοι που εμποδίζουν τους κατασκευαστές να μιλήσουν για την παρουσία αυτών των συσκευών που μπορεί να τοποθετηθούν νομίμως με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν καθαροί, καθαρά τεχνικοί λόγοι για τις, τους οποίους οι κατασκευαστές δεν μιλάνε για την παρουσία αυτών των συσκευών. Και μια άλλη ερώτηση για την τεχνολογική ουδετερότητα. Στην απάντηση 10 λέτε ότι η εισαγωγή του παράγοντα συμμόρφωσης είναι ένα μέτρο αντίθετο προς την τεχνολογική ουδετερότητα. Πεςτε μου τη γνώμη σας. Δηλαδή η ευρωπαϊκή πολιτική παροχής κινήτρων για τα ντίζελ μπορεί να συμμορφούνται με την ανάγκη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και με την ανάγκη να διατηρήσουμε καθαρό περιβάλλον. Δηλαδή, μήπως είναι τελικά κίνητρα που ευνοούν μια τεχνολογία εις βάρο μια άλλη και δημιουργούν και προβλήματα. Ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σας. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα για να αποκαλύψουν οι κατασκευαστές ότι υπάρχουν αυτές οι συσκευές. Έχει γίνει στις ΗΠΑ. Και δεν έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τους κατασκευαστές. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Το ερώτημά σας για την ε, τεχνολογική ουδετερότητα ε, δεν ενδιαφέρουσα. Ε, τα πρότυπα Euro 6 δεν είναι τεχνολογικά ουδέτερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα οξύδια του αζότου και τα όρια εκπομπών για τα διζελοκίνητα ε, είναι λιγάκι, τα επίπεδα το, αυτά είναι λιγάκι υψηλότερα για τους διζελοκινητές από ότι για τους βενζελοκίνητες. Αν χρησιμοποιήσετε τον ίδιο παράγοντα συμμόρφωσης σε διαφορετικά αυτά, καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα και πάλι έχετε το όριο για το δίζελ. Ο παράγοντας συμμόρφωσης. Το χρειάζονται οι δισελοκινητήρες, γιατί οι πραγματικές επιδόσεις τους σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης δεν είναι τόσο καλές όσο των βενζινοκινητήρων. Υπάρχει ένα αντεπιχείρημα όμως που δεν αφορά τι εκπομπέ οξυδίου του άνθρακα, αλλά ε, των σωματιδιακών ρήπων. Έχουμε ένα υποσύνολο ε, βενζινοκινητήρων που μπορεί όχι να έχουν πρόβλημα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, θα πρέπει να το δούμε αυτό του επόμενους μήνες ή χρόνια. Και τα RDE είναι προορατικές ε, εκπομπές και θα μα βοηθήσουν τόσο ώστε να περιορίσουμε του σωματιδιακού ρήπου για να μην φτάσουν στο επίπεδο που έχουν φτάσει σήμερα ε, οι ρήποι που είναι τα οξύδια του αζότου δηλαδή. Πάμε τώρα στον ε, δεύτερο γύρο. Τρία λεφτά στον καθένα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φράγκο, ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Θα ήθελα να επανέλθω στο γράφημα της παρουσίασής σας, στη σελίδα 5. Και την τεχνολογία CR. E Και την υπόθεση BMW G23. 320. Υπάρχουν διάφορε τεχνολογίες, αν δει κανεί το γράφημα βεβαίω. Υπάρχουν διάφορα αυτοκίνητα με την ίδια τεχνολογία και παρόλα αυτά καταλήγουν σε διαφορετικές επιδόσεις εντελώς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, η τεχνολογία CR είναι μια ενεργή τεχνολογία. Πρέπει κανείς να να, πρέπει να την διαχειρίζεται η ECU του, ε, του οχήματος. Ε, εξαρτάται δηλαδή από την χρήση, από την εφαρμογή της τεχνολογίας. Κάποια ε, αυτοκίνητα μπορούν και κάνουν, παίρνουν καλές αποφάσεις και έτσι κρατούν χαμηλές τις ε, εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου, αλλά εξαρτάται πάντοτε και από τις συνθήκες ε, οδήγησης. Τα, τα στοιχεία αυτά προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, σε διαφορετικές συνθήκες, σε διαφορετικούς χώρους έγιναν οι δοκιμές υπό διαφορετικέ συνθήκες, οπότε ε, δεν, είναι, δεν θα ήταν λογικό ε, όλα τα οχήματα ΙΣΑ να ε, συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Λέτε όμως ότι εξαρτάται και από την ποιότητα αυτής της τεχνολογίας για το αν αποτελεί ενσωματωμένο εξοπλισμό ή αν έχει ε, προέλθει από άλλον ε, προμηθευτή. Ε, εξαρτάται και από το, όχι τόσο από το software όσο από το hardware και από διάφορους άλλους παράγοντες. Είναι δύσκολο κανείς να, ε, να ε, συνυπολογίσει και να πάρει τα ίδια αποτελέσματα ακόμα και όταν ε, μιλούμε για, το, για έλεγχο δύο φορές στο ίδιο αυτοκίνητο. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να συνδυαστεί το hardware με το software και έτσι οι αυτοκιν κάποιες ε, αυτοκινητοβιομηχανίες είναι καλύτερες στο συνδυασμό του software και του hardware από ότι κάποιες άλλες. Αυτό προκύπτει. Ναι, είναι μια λογική εξήγηση αυτή που δίνεται ε, για τις διαφορές. Εξηγεί σε μεγάλο βαθμό, εν πάση ε, αυτή τη διαφορά στα αποτελέσματα. Αποτελεί έναν ε, συνδυασμό και των δύο, αλλά σίγουρα το λογισμιακό ε, το λογισμικό παίζει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να έχει κανείς το καλύτερο hardware στον κόσμο, αλλά αν δεν συνοδεύεται από ένα καλό λογισμικό, τότε τα αποτελέσματα που θα πάρει δεν είναι καλά. Ναι, μιλάμε πάντοτε για δεδομένα μίας ώρας. Κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Καθλίν, ευχαριστώ κύριε Φράγκο. Όπως γνωρίζετε, 400.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της ρήπανσης του αέρα. Ε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την πολιτική. Ποιες διαδικασίες που έχουν υιοθετήσει η ΕΠΑ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εσείς ε, σε ποιες συνθήκες ε, προτείνεται να γίνονται οι δοκιμές των, των οχημάτων. Ε, είπατε κάποια πράγματα, αλλά τι θεωρείτε εσείς ότι είναι οι τρεις βασικότερες προτεραιότητες για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Πρόκειται για ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας και καλό είναι να μην το ξεχνάμε. Γιατί θέλουμε καθαρό αέρα και όχι μόνο στα εργαστήρια εκπομπών, αλλά και στις πόλεις μας προφανώς. Υπάρχουν στοιχεία της Αμερικανικής νομοθεσίας που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ένα ζήτημα το ανέφερα ήδη νωρίτερα και αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης και τους ορισμούς του πότε κανείς μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτική βαθμονόμηση και πότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο και αυτό όσον αφορά και τα συστήματα αναστολής. Ε, ένα άλλο στοιχείο που λείπει από το αμερικανό, αμερικανικό πλαίσιο είναι η έλλειψη PEMS στην έγκριση τύπου. Άρα κανένα σύστημα δεν είναι άψογο και έχει κάποιες, κάθε σύστημα έχει κάποιες ε, ελλείψεις. Χρειάζεται ωστόσο να επενέσουμε τα θετικά στοιχεία του κάθε συστήματος και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ΙΠΑ έχουν ένα πιο στιβαρό σύστημα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επικεντρώνονται στην ε, συμμόρφωση ε, στο στάδιο του σέρβις, κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη αλλά ελπίζουμε να υιοθετηθεί ε, με την ευκαιρία του, του νέου, ε, της νέας πρότασης για το πλαίσιο ε, έγκρισης τύπου. Η πρώτη μας ε, σύσταση είναι να ενσωματωθεί το RDE στην συμμόρφωση στο στάδιο του service. Οι διαδικασίες υπάρχουν ήδη, άρα θα είναι σχετικά εύκολο να επεκτείνουμε αυτήν τη δοκιμή προκειμένου να καλύπτονται πλέον και οχήματα που βρίσκονται ήδη σε χρήση και κάτι τέτοιο θα είναι πολύ θετικό βήμα. Επίσης προτείνουμε οι συντελεστές συμμόρφωσης να μειωθούν προκειμένου να ανταποκρίνονται και να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της τεχνολογίας, της τεχνολογίας ώστε να ε, δοθούν και κίνητρα για την υιοθέτηση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών και θα θέλαμε και να επεκταθούν οι οριακές συνθήκες της δοκιμής RDE προκειμένου να ε, καλύπτεται η ευρύτατη γκάμα πραγματικών συνθήκων ε, οδήγησης. Κύριε Συντομότατα. Να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Ζάλμπα Καταρχάς, το ICCT κινείται αυτόνομα, κάνει δικές της επαληθεύσεις. Στις 13 Νοεμβρίου του 2015, σε μια γερμανική εφημερίδα όμως, δημοσιεύτηκε μια είδηση ότι το 2011 κάποιοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσαν το ICCT για κάποιες διαφορές ε, στις εκπομπές και ζήτησαν μια δράση για να καταγγελθεί η αδράνεια της Κομισιόν. Οι πάλι της Κομισιόν το κάνουν αυτό, έτσι. Αυτό μας είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Θα ήθελα να το σχολιάσετε παρακαλώ αυτό το στοιχείο, αυτή την είδηση που όλοι ξέρουμε. Δεύτερο, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Ζάρμπα. Η ICCT το 2014 μίλησε καλά για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση για το πώς κάνει αυτές τις δοκιμές για τις ε, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες. Ε, και σε μια άλλη δήλωση πιο πρόσφατη του Δεκεμβρίου του 2015 της ICCT έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκαπανέας στη χρήση ε, πραγματικών, ε, δηλαδή μέτρηση των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Την επένεσε λοιπόν. Σχολιάστε το παρακαλώ και αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο. Η ICCT Μάλλον, ε, το Πανεπιστήμιο της ε, Δυτικής ε, Βιρτζίνια ζήτησε να διερευνηθεί το θέμα των εκπομπών των δισελοκινητήρων. Γιατί ζήτησε τέτοιες, τέτοια στοιχεία η ICCT ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Βιρτζίνια να, κάνει, να διερευνήσει το θέμα αυτών των εκπομπών. Εάν μιλάτε για δύο... Κάτι για δύο λεφτά, σας μένει ένα λεφτό μόνο, έξτρα. Δεν το ξέρω αυτό το άρθρο στο... στη γερμανική εφημερίδα και δεν δούλευα το 2012 στο ICT. Και δεν ξέρω ότι ενημερώθηκα ε, το ICCT από υπαλλήλους της Κομισιόν ότι κάτι τρέχει. Α, τον Νοέμβριο 2015. Δεν το ξέρω, δεν το ήξερα. Πιστεύω δεν είναι αλήθεια αυτό. Σας το λέω ειλικρινά. Η ICCT κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάτι, είπατε κάτι τέτοιο. No, so we, we... Α, τους επενέσαμε. Και επιμένουμε στον έπαιρνο αυτό. Ήταν το περιεχόμενο της... Εγώ μιλάω για το περιεχόμενο της καταγγελίας κάποιων υπαλλήλων της Κομισιόν, έτσι. 20 δευτερόλεπτα θα δώσω να απαντήσω. Ο λόγος για τον οποίο ερευνήσαμε τις εκπομπές της Λονοκίνητρας της ΕΠΑ είναι γιατί τότε κάναμε λάθος. Πιστεύαμε ότι το αμερικανικό σύστημα ήταν καλύτερο και ότι δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη για μέτρηση των εκπομπών στις πραγματικές συνθήκες. Πιστεύαμε ότι η αγορά των διζελοκινητήρων ήταν θαυμάσια, η αγορά στην Αμερική, έτσι, και θα, αποδείχ... θα αποδεικνύαμε, ας πούμε, στους Ευρωπαίους ότι είναι καθαροί οι διζελοκινητήρες στην Αμερική. Στην πραγματικότητα όμως δύο από τα τρία αυτοκίνητα με δίζελ κινητήρες στην Αμερική δεν είναι καθόλου καθαρά. Äh, Ευχαριστώ. Είπατε στις γραπτές απαντήσεις σας κύριε Φράγκο ότι οι δοκιμές PEMS όσον αφορά την αξιοπιστία τους ε, είναι πλέον συγκρίσιμες με τις εργαστηριακές μετρήσεις, κάτι όμως που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Σε αυτό προσθέτει το γεγονός ότι οι επικριτές λένε ότι οι τεχνικές διαφορές στα ε, όργανα ΠΕΜΣ είναι προβληματικό στοιχείο και άρα η συγκρισιμότητα είναι δύσκολη. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τη μεθοδολογία και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και ποιες είναι οι εξελίξεις που περιμένετε όσον αφορά την αξιοπιστία των PEM test που θα αναπτύξουν οι κατασκευαστές τα επόμενα χρόνια. I'm sorry. Uh, τα συστήματα PEMS ε, έχουν αποτελέσματα τα οποία μπορούν να... Μάλλον είναι δοκιμές οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν αλλά χωρίς να πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα κάθε φορά. Για ποιο λόγο. Ε, ε, αν έχουμε ένα φορτηγό το οποίο δοκιμάζουμε δύο-τρεις φορές με τον ίδιο κύκλο θα πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα μόνο υπό την ε, προϋπόθεση ότι όλοι οι παράγοντες, οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σταθεροί. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ε, υπάρχουν παράγοντες στους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε στον δρόμο, η κίνηση για παράδειγμα. Ε, σε πραγματικές συνθήκες δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα. Μπορούμε να επαναλάβουμε το πείραμα με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα. Α, δεν έχει όμως σημασία αυτό επιστημονικά. Τα πέμπτα βελτιωθούν σύντομα ήδη έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τα πρώτα που είχαν βγει. Τα πιο πρόσφατα φορητά στήματα μέτρηση εκπομπών είναι και μικρότερα και πιο όμορφα μπορώ να πω. Οπότε και εκεί θα λειτουργήσουν οι δυνάμεις της αγοράς και τα όργανα μας θα βελτιωθούν. Και μάλιστα σύντομα. βέβαια πρωτοστατούντο τις πρωτοστατούσεις αυτής της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Θα μιλήσω γερμανικά. Βάλτε λίγο τα ακουστικά σας παρακαλώ. Δύο ερωτήματα έχω. Οι πετρελαϊκές βιομηχανίες ε, ισχυρίζονται ε, και κάνουν, διαφημίζουν τις ε, διαφορετικές, τη διαφορετική ποιότητα των δικών τους προϊόντων. Εσείς ε, έχετε διαπιστώσει ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Αν ήσασταν βουλευτής, είπατε ότι θα θέλατε περισσότερη πολιτική υποστήριξη. Τι ακριβώς θα προτείνατε όμως. Uh, thank you for your Δεν είμαι ειδικό στα καύσιμα, έτσι να το πω εξ αρχής. Όμως, ίσως θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορές στο προφίλ εκπομπών οξυδίων του αζότου αν το τροφοδοτούσαν με δύο διαφορετικά καύσιμα, αλλά οι διαφορές δεν θα ήταν πολύ μεγάλες. Γιατί, γιατί το άζωτο το οποίο περιέχεται ε, δεν είναι παρόν στα καύσιμα αλλά στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οπότε Οποιασδήποτε διαφορές και αν παρουσιαστούν, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο σημαντικές ώστε ορισμένα καύσιμα να τα θεωρούμε καλά και άλλα χειρότερα σε ό,τι αφορά τα οξύδια του αζότου. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ε, αποφασιστική σημασία παράγοντας. Οπότε δεν θα είχα να κάνω οποιαδήποτε σύσταση για αυτό το ζήτημα. πολιτικές συστάσεις εγώ ζήτησα, όχι για τον ντίζελ. Ε, ίσως δεν κατάλαβα την ερώτησή σας, ε, λέει ο κ. Φράγκο. Ε, ζητήσατε περισσότερη πολιτική στήριξη, έτσι δεν είναι. Στην έκθεσή σας το λέτε αυτό. Οπότε, αν ήσασταν ευρωβουλευτής, εσείς τι θα προτείνατε, ο κ. Φράγκο. Ήδη υπάρχει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας ικανοποιεί αλλά δεν ξέρουμε αν ο τελικός κανονισμός θα ευθυγραμμιστεί με την, πρόταση, την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύουμε μάλιστα ότι η πρόταση της Κομισιόν θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο φιλόδοξη. Αλλά πάντως είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας. Ο κ. Σούλτς. Ευχαριστούμε που πάντα στα ερωτήματά σας. Εγώ είμαι μηχανικός και κάποιες φορές αναρωτιέμαι πώς ερμηνεύει κανείς τέτοιες μελέτες. Νομίζω ότι σήμερα κατάλαβα και αναφέρομαι στο πόρισμα της σελίδας 5 ότι κάτι τέτοιο δεν επαναλαμβάνεται. Δεν, είναι, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής. Ε, ακριβώς επειδή ε, εξαρτάται το απόρισμα από διάφορους παράγοντες. Λέτε δηλαδή ότι ακόμη και αν προσπαθήσει κανείς να επαναλάβει ακριβώς την ίδια δοκιμή δεν θα πάρει τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι αν επαναληφθεί μια μελέτη θα καταλήξετε σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, σε εντελώς διαφορετικά από αυτά στα οποία καταλήξατε την πρώτη φορά θα δώσω την ίδια απάντηση που έδωσα πριν. Ε, η αναπαραγωγή των δοκιμών με PEMS ε, δεν είναι παρόμοια με αυτή των εστιακών δοκιμών. Ε, αυτό μπορεί να το αντιληφθείτε ως αδυναμία της τεχνικής. Αλλά εγώ το βλέπω ως ισχυρό χαρτί, ατού. Γιατί, Γιατί τα PEMS μας δίνουν μια πολύ πλούσια εικόνα του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αν κάθε φορά που έτρεχα την ίδια δοκιμή έπαιρναν το ίδιο αποτέλεσμα, θα ήταν περιορισμένη η αξία της δοκιμής. Ε, και να σας πω κάτι, μακάρι ε, να ε, μου έδινε τα ίδια αποτέλεσμα η δοκιμή κάθε φορά που έτρεχα το πείραμα, γιατί έτσι θα αξιολογούσαμε πολύ πιο εύκολα την συμμόρφωση των αυτοκινήτων. Όμως πιστεύω ότι τα ΠΡΕΜΣ μπορούν να μας βοηθήσουν εξαιτία του πλούτου των πληροφοριών που μας δίνουν. Ευχαριστώ. Δεύτερο ερώτημα, διαφορετικής φύσης. Εσείς, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του κινητήρα. Όσον αφορά την μείωση των εκπομπών, την απόδοση των κινητήρων, πιστεύετε ότι έχουν εξαντληθεί ήδη οι δυνατότητε ή υπάρχουν και περιθώρια βελτίωση. Έχετε κάνει καθόλου έρευνα για αυτά τα ζητήματα τα τελευταία χρόνια ή μήνε. Σαφώς, ε, Σαφώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Οι μηχανές εσωτερικής ε, κάψης ε, δεν έχουν σταματήσει να μας εκπλήσουν εμάς τους μηχανικούς. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και για του βενζινοκινητήρε και για τους πετρελοκινητήρε. Έχουμε πολλές ε, τεχνολογικές ε, δυνατότητες, δρόμους, μονοπάτια τα οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Έτσι ώστε να συμμορφωθούμε τους στόχους διοξιδίου του, διοξιδίου του άνθρακα. Δεν εννοούσα μείωση του βάρους του οχήματος. Μιλώ για τον κινητήρα και την τεχνολογία του κινητήρα. Ναι, η μείωση του βάρους του αυτοκινήτου με ελαφρότερα υλικά αλλά με τον ίδιο βαθμό ασφάλειας ε, θα ήταν ένας πραγματικά πολύ καλός τρόπος να μειώσουμε τις εκπομπές. Θα χρειαζόμασταν μικρότερους κινητήρες. Είναι πραγματικά μια λύση την οποία πραγματικά προτιμούμε. Δεν είναι απαραίτητο όλες οι βελτιώσεις να γίνονται σε επίπεδο κινητήρα. Έχουμε τρομακτικές δυνατότητες καινοτομίας εδώ πέρα. Ο κύριος Έρτουκ. Ευχαριστώ. Ακούσατε σίγουρα και την παρουσίαση από το JRC και ε, θα ακούσατε βεβαίως ότι διαπιστώθηκαν ε, οι μεγάλες διαφορές ε, αλλά παρόλα αυτά ε, είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο χρήση συσκευών αλλίωσης. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξή. Θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί τα αίτια των διαφορών αυτών σε μεγαλύτερο βάθος, πιστεύετε εσείς. Να επανέλθω στο προηγούμενο σημείο για τον ε, χρονισμό και την εισαγωγή του Euro 6. Νομίζω ότι το JRC δεν μέτρησε πολλά οχήματα Euro 6. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο Euro 6. Το ότι τα οχήματα του Euro 5 είχαν ε, κακές επιδόσεις ήταν γνωστό και έτσι είχαν ε, ε, εναποτεθεί πολλές ελπίδες στο Euro 6 για να λυθούν τα προβλήματα. Όταν λοιπόν το JRC έκανε δοκιμές σε οχήματα Euro 5 και έβλεπαν 300 μιλιγκράμμ ε, ανά χιλιόμετρα για παράδειγμα, η αναλογία αυτών των ε, αποτελεσματα αυτών των εκπομπών δεν ήταν ιδιαίτερα κακό ούτε για το Euro 5 ούτε για το Euro 6. Αυτό που όμως επιδίνωσε την κατάσταση είναι το γεγονός ότι οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ υψηλές για το Euro 6. Από 180 mg πήγε στα 80 mg ανά χιλιόμετρο. Άρα τα οχήματα αυτά αναμενόταν ότι θα έχουν ε, ε, εξαιρετικά καλές επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές τους και το γεγονός ότι αυτό δεν ε, υλοποιήθηκε τελικά ε, η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην προσδοκία και στην πραγματική ε, επίδοση των οχημάτων περιγράφει και την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Πάντως δεν είναι πολλά τα οχήματα Euro 6 που έχουν δοκιμαστεί. Ε, ναι ή όχι λέει ο κύριος Έρτουγκ, δεν χρειάζεται να μου ξαναπεριγράψετε την κατάσταση, την ξέρω. Ναι ή όχι. Τι πιστεύετε. Μπορείτε τότε να επαναλάβετε το ερώτημα. Θεωρείτε ότι με βάση τα αποτελέσματα που είχαν υπάρξει θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος τα αίτια που οδήγησαν στα εν λόγω αποτελέσματα. Ναι, Ίσως κατά πάσα πιθανότητα, αλλά το εξετάζεται το ζήτημα με τα μάτια και τις γνώσεις που έχουμε το 2015 και οι μετρήσεις αυτές ε, ξεκίνησαν επί Euro 5 όταν οι γνώσεις μας ήταν ε, λιγότερες. Οπότε ναι, η απάντηση μου είναι ναι, αλλά οι γνώσεις που είχαμε, ε, κάτι τέτοιο δεν ήταν τόσο αυτονόητο όσο φαίνεται ίσως σήμερα. Κύριος Έρτουγκ, θεωρείτε ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να είχε αναθέσει διερεύνηση της υπόθεσης σε κάποιον και συγκεκριμένα στο Κοινό Κέντρο Έρευνας, γιατί είναι προφανές ότι υπήρχαν τεράστιες αποκλήσεις. Οι αποκλίσεις μεγάλωσαν με το Euro 6 και με το Euro 5 ήταν ε, υψηλές, αλλά ακριβώς υπήρξαν αυτές οι προσδοκίες ότι το Euro 6 θα έλυνε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Κάτι που δεν ευωδόθηκε όμως. Με εκπλήσετε κύριε, κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γκυρμπράντη, δεν είχα κάτι να ρωτήσω. Ε, κυρία Γκρόστατ, έχουμε κουραστεί όλοι. Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ αυτοκινήτων του ίδιου μοντέλου που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός και στην Αμερικανική αγορά αφετέρου. Υπάρχουν τεχνολογικές διαφορές σημαντικέ ε, σημαντικές στο ίδιο μοντέλο ανάλογα με το που πωλείται. Ε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσαρμόζουν τα μοντέλα τους ανάλογα με τις αγορές στις οποίες πολλούν. Και δεύτερον, ποια είναι η σχέση που έχετε αυτή τη στιγμή με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τώρα σε σχέση με την περίοδο πριν την αποκάλυψη του σκανδάλου. Thank you for your So... Απάντηση. Το Σεπτέμβριο του 2015 πριν το σκάνδαλο είχαμε δημοσιεύσει μια έκθεση που εξέταζε τις ε, τεχνολογίες ε, ελέγχου εκπομπών σε αυτοκίνητα με πετρελοκινητήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ και είδαμε σημαντικές διαφορές. Τα αποτελέσματα με δύο λόγια ήταν ότι η, τα συστήματα LNT στην Ευρώπη ε, παγίδων οξυδίου του αζότου ήταν ε, πιο διαδεδομένα και είχαν αυξήσει το μερίδιο της αγοράς τους από το 2012 στο 2014. Αντιθέτως, ε, στις Πολιτείες χρησιμοποιείται πιο πολύ η ε, τεχνολογία NCR. Ε, η BMW από την άλλη μεριά ε, από το 2014 και μετά ξεκίνησαν να παράγουν όλα τους τα αυτοκίνητα με δύο τεχνολογίες SCR και LNT ε, με δύο τεχνολογίες δηλαδή, ενώ όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, στον, και στις Ηνωμένες έχουν μόνο μία τεχνολογία. Δεν προσπαθώ να το κρίνω αυτό, απλά πιστεύω ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται στην ύπαρξη πιο αυστηρών κανόνων και προδιαγραφών στις ΗΠΑ. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσαρμόζονται στα αυστηρότερα στάνταρ, στα αυστηρότερες προδιαγραφές και κάνουν περισσότερες ε, προσπάθειες ε, ε, εφαρμογής της ερευνάς τους σε συγκεκριμένες αγορές. Όταν είναι πιο αυστηροί οι κανόνες, η τεχνολογία προχωράει πιο γρήγορα και ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο αυστηρή. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Ε, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα και είμαστε και πιο αισιόδοξοι για το μέλλον μετά από αυτήν. Μια και όμως συζητούμε κάτι το οποίο το δημοσίευσατε εσείς, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ε, αν τα συμπεράσματά σας σημαίνουν ότι η ενδεχόμενη απάτη ε, περιορίζεται στη Volkswagen και στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ή αν παρόμοια συμπεριφορά θα μπορούσαν να έχουν δείξει και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ε, ο κ. Φρανκό, δεν μπορούμε εμείς με βάση τα στοιχεία που έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε πει. Ότι δηλαδή δείχνει να υφίσταται ένα γενικευμένο πρόβλημα μετρήσεων εκπομπών για τα αυτοκίνητα ε, με πετρελοκινητήρες γύρω 6. Αν αυτό έχει σχέση με την ε, χρησιμοποίηση διατάξεων παράκαμψη όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Εσείς πιστεύετε ότι ε, ορισμένοι, ορισμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, μάλλον οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πιο επιρρεπείς στη χρήση τέτοιων ε, διατάξεων. Η απάντηση. Οι τεχνολογίες είναι διαθέσιμες σε, όλους και ο καθένας κάνει τις επιλογές του με βάση τους δικούς του περιορισμούς, ε, κανονιστικούς, οικονομικούς κλπ. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι ε, έχουμε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες στους οποίους δεν ελέγχουμε και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το την πηγή αυτών των διαφορών. Στο, στην Ευρώπη τι είναι πιο σημαντικό, το κανονιστικό πλαίσιο, η τεχνολογία, η διαθέσιμη τεχνολογία, είναι το γεγονός ότι ε, από οικονομικής πλευράς ευνοούνται κάποιες επιλογές εναντί άλλων. Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές δεν, δίνουν, είναι τόσο πολύ ευαισθητοποιημένοι στην Ευρώπη σε σχέση με το περιβάλλον. Ε, πολύ ωραίες οι μελέτες και μαθαίνουμε πολλά για σας. Υπάρχει ένα προφίλ στην Ευρώπη όχι, σίγουρα δεν είναι οι καταναλωτές. Ε? Οι καταναλωτές δεν κάνουν ε, συγκεκριμένες επιλογές τεχνολογίας. Ε, ένα οχήμα το οποίο έχει πιστοποιηθεί ως Euro 6 θεωρείται καθαρό. Οπότε οι καταναλωτές δεν κάνουν διάκριση ε, ανάμεσα σε ένα καθαρό και ένα βρώμικο διζελοκινητήρα δεν έχουν τις πληροφορίες για να το κάνουν αυτό. Ε, αυτή, ε, αυτή η επιλογή γίνεται από τους ίδιους τους κατασκευαστές. Κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ κύριε Φράγκο για την εκθεσή σας. Πολύ γρήγορα. Πιστεύετε ότι αυτό που λείπει στην Ευρώπη είναι αυτό που έχουν οι ΗΠΑ, αυτή η υπηρεσία δηλαδή που είναι ανεξάρτητη, που έχει εξουσία, που έχει πόρους και που επιτρέπει με απεριόριστες εξουσίες να αλλάξει τα δεδομένα έστω και απότομα. Δεν πιστεύετε ότι στην Ευρώπη σήμερα θα χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχων πραγματικά ανεξάρτητη και που θα μπορούσε να επαληθεύει τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Και παράλληλα να αλλάξει το πλαίσιο ή να δώσει έτσι μια θετική όθηση, ας πούμε, στην αυτοκινητοβιομηχανία και να την εξαναγκάσει, αν θέλετε, με ένα καλό momentum να σεβαστεί τους κανόνες. Ομοθυμαδών θα απαντούσαν ε, στο ICCT, ναι. Σίγουρα μια ευρωπαϊκή υπηρεσία χρειάζεται τέτοιου τύπου. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό βέβαια είναι εφικτό ή ρεαλιστικό να υπάρξει κάτι τέτοιο, να δημιουργηθεί μια τέτοια υπηρεσία. Γιατί υπάρχουν 28 διαδικασίες έγκρισης τύπου στην Ευρώπη σήμερα. Και πολιτικός πώς θέλει, χρειάζεται πραγματικά και θέληση και πολλά κίνητρα για να ξεφορτωθούμε τις 28 διαφορετικές διαδικασίες και να, τις, ε, και να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος. Ανταυτού η Κομισιόν προτείνει κάτι ε, αντίστοιχο να εστιάσουμε στην αρμόνιση και ο ρόλος της ε, εποπτείας να αναβληθεί, να αναλυθεί από εκεί, από αυτήν, κρατώντας όμως τις ε, διάφορες υπηρεσίες. Μπορεί να είναι μια ενδιάμεση λύση για να έχουμε κάποιες από, τις, ε, τα θετικά και από τα πλάσα ας πούμε, των Αμερικανών, δια, διατηρώντας όμως και τις ευρωπαϊκές δομές. Αλλά εντάξει, αυτό το μέλλον θα το δείξει. Προηγουμένως είπατε ότι δεν πιστεύετε πολύ στο καθαρό ντίζελ. Έτσι, για να παίξουμε λίγο πινκ-πονγκ τώρα. Ούτε εγώ πιστεύω. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την ταύτιση απόψεων. Δεν πιστεύετε ότι για αυτό το θέμα σήμερα η εστίαση θα πρέπει να δοθεί στη δημόσια υγεία των πολιτών δηλαδή και να πούμε συγκεκριμένα ότι η υπηρεσία αυτή θα έχει αυτό το ρόλο Δηλαδή, να κάνουμε εστίαση στην δημόσια υγεία όπως κάνουν και οι Αμερικανοί. Η εντολή της Αμερικανικής Προστασία του Περιβάλλοντο είναι ακριβώς να προστατεύει και το περιβάλλον και την υγεία των Αμερικανών πολιτών. Και το κάνουμε πολύ καλά. Ξέχασα το πρώτο τη ερώτηση. Είμαι σίγουρος ότι είχα την απάντηση. Κουραστήκαμε, λέει η Πρόεδρος, όλοι μας. Είναι 6.30 συνάδελφοι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση, πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Φράνκο για τις μακροσκελείς σας απαντήσεις. Αν οι συνάδελφοι έχουν και άλλες ερωτήσεις προς τα ICCT, μπορούν να τις υποβάλουν γραπτός. Και μην ανησυχείτε, θα εξασφαλίσουμε απαντήσεις. Υπάρχουν και τα πρακτικά στα αγγλικά. Θα υπάρχουν μάλλον στα, σε 10 μέρες. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 28 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ.